Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ελληνικού Συνεδρίου, ευρωβουλευτές, συνεργάτες και λοιποί συμμετέχοντες στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αντιλαμβάνω εγώ την Προεδρία σε αυτή τη συνεδρίαση, γιατί ο κύριος Μαγκίστρης, ο, ο πρόεδρος είναι άρρωστος. Ίσως μπορέσει αύριο να έρθει. Αλλά δεν είναι βέβαιο. Πάντως απόψε τον αντικαθιστώ εγώ. Έχετε λάβει πιστεύω το κοκομπιού εμφού και τα έγγραφα συνεδριάσεως με την ημερήσια διάταξη η οποία μένει χωρίς ε, αλλαγές. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζητούν κάποιες μικρές τροποποίησεις. Σας παραπέμπω λοιπόν στην ημερησία διάταξη, προ... Ε, έγκριση πρακτικών, ανακοινώσεις του Προέδρου, έκθεση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με τον κύριο Τόμας Ντόιτς. Και μετά έχουμε την ειδική έκθεση 2000, ε, υπαριθμών 10-2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για ειδικά μέτρα για την Γεωργία με την κυρία Κέστιγκερ. Στο σημείο 6 6-Δ άρνηση απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ΣΕΠΟΛ. Οι σοσιαλιστές δημοκράτες ζητούν το σημείο 6 να έρθει πριν από το υπαριθμόν 5. Ε, ζητούμε φυσικά και τη γνώμη των εισηγητών, της κυρίας Ματσιού και της κυρίας Κρέστιγκερ, εάν δεν έχουν αντίρρηση, μπορεί να γίνει δεκτή η τροποποίηση αυτή. Κύριε Γκάιερ, εντάξει είμαστε. Πολύ καλά. Τροποποιεί τη μερίσια διάταξη, εάν δεν έχουν αντίρρηση οι δύο συνάδελφοι. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου του 2010 που έχετε λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις προς τα πρακτικά. Εγκρίνονται. Εάν έχουν, παρακαλώ να μας τις κοινοποιήσετε. Ανακοινώστε το Πρόεδρο. Δεν έχουμε τίποτε το ιδιαίτερο. Έχετε στο έγγραφο Κοκομπιού Info τις γλώσσες. Έχουμε την αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου της συνεδρίασής μας. Μην ξεχνάτε ότι όποιο πατάει το μικρόφωνο στρέφει, στρέφει και την κάμερα πάνω του και μαγνητοσκοπείται. Μην ξεχνάτε λοιπόν να χαμογελάτε. Και ε, για το σημείο ε, της αυριανής συνεδρίας του που αφορά το ελεγκτικό συνεδρίο, ο κύριο Γκαλέα δεν θα είναι παρόν, αλλά η κυρία Μποσί ο κύριος Όση ε, μέρος του ενεκτικού Συνεδρίου. Η αλλαγή οφείλεται σε λόγους υγείας. Αυτά λοιπόν. Όπως είπαμε, ο κύριος Γκαλεά ε, θα απουσιάζει και θα αντικατασταθεί από τον κύριο Όση. Περνώ λοιπόν τώρα στην... Ε, ειδική έκθεση παριθμών 2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα διευθυντικά μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε ω προ την προμήθεια σε είδωρ για οικιακή κατανάλωση. Η ομάδα του κυρίου Μάσιμο Βάρη έχει ετοιμάσει την έκθεση, ο κύριος Ντόιτς είναι εισηγητής και ως εκ τούτου προτείνω πρώτα να ακούσουμε τι έχει να πει το ελεγκτικό συνέδριο και στη συνέχεια τον κύριο Ντόιτς και τους λοιπούς συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Βάρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ειδική έκθεση που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αντικείμενο την χρηματοδότηση για την υλοποίηση υποδομών στον τομέα της ε, παροχής ε, νερού για οικιακή χρήση. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εντάσσεται στην γενικότερη περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης που όπως γνωρίζουμε ε, προβλέπει την προγραμματισμένη χρήση των, ειδικών, των φυσικών πόρων με βάση την ανάπτυξη των βιώσιμων πόρων. Ε, η ειδική έκθεση λοιπόν σχετίζεται με τους ευρωπαϊκούς πόρους που, που στόχο έχουν την υδροδότηση για οικιακή χρήση και να δούμε αν αυτοί οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε εξετάσει τις καλύτερες λύσεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, των ε, ενδιαφερομένων περιοχών. Αν όντως ε, τα έργα που γίνονται αφορούν την υδροδότηση για γεωργική χρήση και αν έγιναν σύμφωνα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μιλάμε για τέσσερα κράτη-μέλη, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία που πήραν περίπου το 90% της ευρωπαϊκής οικονομικής στήριξης για την περίοδο 2000 με 2006, σύνολο περίπου 4 δις ευρώ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ε, βασίζονται σε μια άμεση εξέταση ενός δείγματος 29 προγραμμάτων που έχουν ε, ολοκληρωθεί. Το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι το εξής η ευρωπαϊκή δαπάνη που στο έχω είχε την συγχρηματοδότηση δομών, υποδομών μάλλον υδροδότησης συνέβαλε στη βελτίωση του νερού για οικιακή χρήση, αλλά θα μπορούσαν να είχαν και καλύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όμως, είναι, Ποια είναι λεπτομερώς τα βασικά στοιχεία που εκτίθενται σε αυτή την έκθεση όσον αφορά την επιλογή λύσεων που στόχο έχουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι στην ανάλυση των προπολογισμών συχνά δεν λήφθη υπόψη η τάση για μείωση της κατακεφαλής κατανάλωσης πόσιμου ύδατος και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των πόρων που ήδη ήταν διαθέσιμοι. Επιπλέον ακολουθήθηκε κατά κύριο λόγο μία προσέγγιση του τύπου supply side, δηλαδή με προσανατολισμό να αυξηθεί η προσφορά. Πράγμα το οποίο ευνόησε την δημιουργία υποδομών που στόχο έχουν την εκμετάλλευση επιπλέον πόρων αντί να ακολουθηθεί μία προσέγγιση βιώσιμου τύπου με βιώσιμης χρήσης που να έχει στόχο την αποτελεσματική χρήση και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος που στόχο θα είχε την περιορισμό των απολειών από το δίκτυο υδροδότησης, βελτίωση των, της χρήσης, δηλαδή μείωση των σπαταλών και η πιο ευέλικτη χρήση των, υπάρχων των υπαρχών διαθέσιμων ε, ε, υποδομών. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ή προγράμματα του Ταμείου Συνοχής. Ε, στις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών όταν ε, στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονταν και τα πιο γενικά επιχειρησιακά προγράμματα επέφεραν μια προστιθέμενη αξία στο θέμα της αξιολόγησης των ετοιμάτων ε, για συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν πολλές φορές έχει συμπεριλάβει όρους για να λάβει την απόφαση της επιχορήγησης, όμως δεν απαλήθευσε πάντοτε επαρκώς την υλοποίηση αυτών των όρων. Το συνέδριο στην ειδική έκθεση λοιπόν έχει διατυπώσει τις εξής συστάσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναγνώριση των διαθέσιμων πόρων και των τάσεων εξέλιξης της ε, κατακεφαλήν κατανάλωσης ε, ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες κάθε περιοχής, να λάβουν υπόψη εναλλακτικέ λύσεις από εκείνες ε, που αφορούν μόνο την προσφορά, να βασιστούν δηλαδή σε μια λογική ε, εκμετάλλευσης ε, που, μάλλον, που βασίζονται στην λογική της εκμετάλλευσης νέων πόρων. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει πριν από την εκχώρηση των κονδυλίων αν στις εν λόγω περιοχές έχουν υιοθετηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτραπεί η επατελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τέτοια, ε, τέτοιο είδος μέτρα. Τώρα, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονταν μέσω της χρηματοδότηση, ο έλεγχο έδειξε πως τα προγράμματα γενικά έφεραν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση του όγκου του διαθέσιμου ύδατος, την κάλυψη από πλευρά του δημοσίου δικτύου υδροδότησης, ποιότητα του νερού και συνέχεια διάρκεια τη υπηρεσία. Ωστόσο, ορισμένε εγκαταστάσεις, αν και έχουν ολοκληρωθεί, δεν είχαν ακόμα τεθεί σε λειτουργία στην εποχή του ελέγχου λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση ή στην έναρξη λειτουργία των συμπληρωματικών υποδομών. Ενώ άλλες εγκαταστάσεις ε, φάνηκε να περιορίζονται από ε, διάφορα προβλήματα που δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστούν. Ε, βρίσκουμε ότι δεν είχαμε αρκετές αποδείξεις σε σχέση με τα αποτελέσματα που επετεύθηκαν. Στη στιγμή δηλαδή που είχαμε αυτές τις πληροφορίες ε, που προέρχονταν από την παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων ήταν μερικές και ελλειπείς αυτές οι πληροφορίες. Η δε δεν έχει πάντοτε παληθεύσει την ε, πραγματοποίηση, την υλοποίηση των έργων. Όσον αφορά τις συστάσεις που ακολουθούν από ε, αυτά τα απορίσματα, το συνέδριο καλεί τα κράτη-μέλη να επαληθεύουν ήδη από τη φάση του προγραμματισμού τις οι συμπληρωματικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων να γίνονται εγκαίρως και να θεσπίσουν πιο αποτελεσματικά μέσα για την παρακολούθηση. Η Κομισιόν από την πλευρά της θα πρέπει να ορίσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των προγραμμάτων και να ακολουθήσει την εφαρμογή των όρων που προβλέπει στις αποφάσεις χρηματοδότησης. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική πτυχή που αντικατοπτρίζεται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις και έξτρα κόστη στην υλοποίηση των προγραμμάτων που βασικά οφείλονται στην, στον ελληπή προγραμματισμό. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των υποδομών που επισκεφθήκαμε, που βασικά μετράται με βάση δύο παραμέτρους, δηλαδή το ποσοστό χρήσης της υποδομής σε σχέση με ε, τις δυνατότητές της και το ποσοστό ύδατος που λόγω των απολειών δεν ε, χρεώνεται, ε, συχνά ήταν περιορισμένη. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη φάση του προγραμματισμού σε παράγοντες που είναι πιθανά, πιθανά αίτια καθυστερήσεων. Να βελτιώσουν την ποιότητα της ανάλυσης επί τη βάση των οποίων ε, ε, βασίζεται το μέγεθος των εγκαταστάσεων, να εξετάζουν συστηματικά τη δυνατότητα μιας προσέγγισης με διαδοχικές φάσεις ώστε να αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις με βάση την εξέλιξη των αναγκών. Τέλος, η διαδικασία καθορισμού της Ευρωπαϊκής Συμβολής που βασίζεται στην ανάλυση κόστους οφέλους που παρουσιάζεται πριν από τα προγράμματα έδειχνε, έδειξε σημαντικές ελλείψεις και δεν εγγυάται την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Μεταξύ άλλων ε, ε, δεν δόθηκε παρκής προσοχή στην γενικότερη δυνατότητα ε, για προγράμματα που θα έδιναν ε, έσοδα, θα οδηγούσαν σε έσοδα και χρέωση των υπηρεσιών έτσι ώστε να μειωθεί το κενό της, ανάμεσα στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος και άρα να διατηρηθεί σε λιγότερο σε χαμηλότερο επίπεδο η ευρωπαϊκή συμβολή. το κόστος μακράς περίοδου, δηλαδή η απόσβεση των εγκαταστάσεων και το περιβαλλοντικό κόστος αγνοείται μέσα στον προγραμματισμό. Τώρα, για τα, τα χαμηλά κόστη δικαιολογούνται μέσω των κοινωνικών αιτίων ε, που σχετίζονται με τα χαμηλά έσοδα ε, των οικογενειών στις συγκεκριμένες περιοχές και αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε πως το κόστος για ε, την υδροδότηση δεν πρέπει να ξεπερνά κάποιο κρίσιμο σημείο για τις ε, οικογένειες εφόσον πρόκειται για βασικές παροχές. Η έκθεση Θεωρεί τέλος ότι η τιμή που χρεώνεται στις οικογένειες θα πρέπει να ορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να λαμβάνει υπόψη το κόστος λειτουργίας αλλά και το κόστος ανανέωσης ανακαίνησης των υποδομών αλλά και να παροτρύνει τη βιώσιμη χρήση του πόρου. Αυτή, αυτές είναι οι αρχές εξάλλου που αναφέρονται στην οδηγία πλαίσιο για το είδωρο που ρητός αναφέρει το ε, ότι το κόστος χρήσης ε, θα, είναι, ε, θα επιβαρύνει τον χρήστη. Αυτή είναι η αρχή η οποία αποτελεί αντικείμενο της σημερινής έκθεσης. Ε, το ηλεκτρικό συνέδριο λοιπόν συστήνει η Κομισιόν να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των, των ε, ε, δημοσιονομικών αναλύσεων που παρουσιάζονται όταν γίνονται τα αιτήματα χρηματοδότησης και να εφαρμόζει πιο αυστηρά την αρχή της ανάκτησης του κόστους. Αυτή είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και σας βεβαίως, αλλά και όλη σας την ομάδα για το εξαιρετική δουλειά σας και τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Ντόιτς κατέγραψε τα όσα περιλαμβάνει η εκθεσή σα και δημοσίευσε την, ε, το έγγραφο εργασίας με τις έξι Τον παρακαλώ λοιπόν τώρα να μας παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις και αν χρειαστεί θα ρωτήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να λάβει το λόγο. Φυσικά και οι συνάδελφοι που το επιθυμούν μπορούν να με ενημερώσουν. Κύριε Ντόιτς, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω τα πρώτα μου σχόλια, για τον αριθμό. Ευχαριστώντας το προσωπικό της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλους τους συναδέλφους και όσους ανέλαβαν την διοργάνωση ε, της σημερινής συνεδρίας, αλλά πάνω απ' όλα την ε, διατύπωση της εκθέσεως επέδου ελεκτικού συνεδρίου. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα ως προς την ε, γαλλική καμπίνα, μάλλον τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Καλώς λοιπόν, ευχαριστώ. Καταρχάς ρωτώ εάν με ακούτε όλοι σε όλες τις γλώσσες. Ακούγομαι καλά. Ξέρουμε ότι γίνεται αναμετάδοση της συνεδρίασης από το διαδίκτυο. Όποιος λοιπόν παρακολουθεί την ε, συνεδρίαση αυτή θα βλέπει μάλλον προς το παρόν μια κενή οθόνη ε, γιατί ανάλογα με το μικρόφωνο το οποίο ανάβει στρέφεται και η κάμερα στο αντίστοιχο κάθισμα. Αν όμως πατήσω εγώ το άλλο μικρόφωνο το οποίο θα ε, προσελκύσει το ενδιαφέρον της, της ε, κάμερας δεν θα ακούγεται η φωνή μου γιατί αυτό το μικρόφωνο φαίνεται δεν δουλεύει. Εν πάση καλύτερα να με ακούτε παρά να με βλέπετε και συνεχίζω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Βάρη, τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, καθώς και ολόκληρη την ομάδα για αυτή την ιδιαίτερα υψηλού επίπεδο έκθεση. Έχουμε λοιπόν ένα έγγραφο, βάσει του οποίου πιστεύω μπορούμε να προβούμε σε μια εις ανταλλαγή απόψεων και διεξοδική συζήτηση. Δεύτερον, δεν θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση με την ευκαιρία αυτή που προσφέρει η ειδική έκθεση. Και βέβαια το έγγραφο εργασία τη Επιτροπή, το οποίο έχω αναλάβει εγώ τη διατύπωση, διότι πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το καθήκον που έχει φορτιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την ε, διαφύλαξη των υδάτινων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερη σημασία βέβαια αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα στην διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ε, υδάτινων αποθεμάτων. Όμως αυτό δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας σήμερα, τουλάχιστον όχι απευθείας. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην ε, διαφύλαξη των υδάτινων πόρων και στα συναφή ζητήματα. Όταν μας απασχολούν ζητήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, η αύξηση της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη. τα αποθέματα σε υδρογονάνθρακες, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ούτω καθεξής και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη ιδιαίτερος η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερος του κ. Βάρη, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στην ουσία τους και να επικεντρωθούμε στη σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, όπως την υπογραμμίζει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και πιστεύω ότι και η έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα σταθεί στα ίδια σημαντικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, όπως επεσήμανε και το ελεγκτικό συνέδριο με του κ. Βάρη, μεταξύ 2000 και 2006, που ήταν η περίοδος ε, ελεγχθή από το συνέδριο, Και θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερως τις ε, τέσσερις χώρες στις οποίες ε, δόθηκε έμφαση Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και θα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι η σημερινή, η τωρινή περίοδος προγραμματισμού, δηλαδή 2007 με 2013, όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη έχουν δικαίωμα οι 15 κράτη-μέλη. Πάντοτε όσον αφορά τα προγράμματα για την πιο βιώσιμη χρήση των ε, υδάτινων πόρων. Μιλάμε για 25 δις για αυτήν την ε, προγραμματική περίοδο. Δεν θέλουμε να ε, μεταβιβάσουμε, να αναπαράγουμε τις εμπειρίες των 10-15 χρόνων που πέρασαν. Όχι. Θέλουμε όμως να μπορέσουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας να φτάσουμε σε συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τα 25 δις που έχουμε στη διάθεσή μας με το πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη των υποδομών. Τώρα, στόχος μου δεν είναι να επαναλάβω όλα όσα μας είπε ο κύριος Βάρη. Ως εισηγητής, συμμερίζομαι απόλυτα τα όσα μας εξέθεσε ως πορίσματα της ανάλυσης. Θα ήθελα να σας ε, Αναφέρω ωστόσο κάποια στοιχεία από τη δική μου έκθεση. Καταρχήν θα ήθελα να υποστηρίξω ακόμα μια φορά ότι δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε τη στρατηγική σημασία του νερού για τον 21ο αιώνα. Ω εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντική η διατήρηση αυτού του φυσικού πόρου που έχει στρατηγική σημασία. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Να πω επίσης ότι στην έκθεσή μου εγώ μιλώ για την ε, ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου και υπογραμμίζω την σημασία για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι αλήθεια ότι μιλάμε πάντα για ολοκλήρωση, για ένταξη. Ένα σωρό χρησιμοποιούμε περίπλοκες φράσεις, αλλά συγκεκριμένα χρειάζεται να αναζητήσουμε τον συνδυασμό της οικονομικής και της περιβαλλοντικής προοπτικής όσον αφορά την εγγύηση της προστασίας των υδάτινων πόρων. Δεν μπορούμε δηλαδή να κατακαιρματίσουμε το θέμα του περιβάλλοντος Εντάξει, μπορεί να μιλάμε για επενδύσεις στις υποδομές ή για διαχείριση και να εστιάζουμε περισσότερο στην οικονομική επιτυχία του θέματος, αλλά δεν μπορούμε να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτό και να βάζουμε στην άκρη όλα τα υπόλοιπα όπως ε, το περιβάλλον, τα θέματα τα περιβαλλοντικά για την συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπε τώρα και ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνεδρίου ότι πρέπει δηλαδή να γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένος και αυστηρός προγραμματισμός. Η σημερινή κατάσταση δεν γίνεται να συνεχιστεί. Ε, προφανώς πρόκειται για πολύ σημαντικό πόρο, άρα λοιπόν όσον αφορά την χρήση του πόρου αυτού, Όταν επενδύουμε ευρωπαϊκά χρήματα για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται συγκεκριμένε αξιολογήσει και συγκεκριμένε προβλέψει καταρχήν. Οι αρχέ ε, διαχείριση δεν έχουν συγκεκριμένη ιδέα. για το σύνολο της κατανάλωσης για την επόμενη περίοδο, δηλαδή την περίοδο για την οποία γίνεται ο προγραμματισμός. Επενδύονται δηλαδή χρήματα, επενδύονται κονδύλια της Ένωσης για να αυξηθεί ο όγκος του καθαρού νερού, του πόσιμου νερού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν προγράμματα για την μείωση της κατανάλωσης. Από τη μια πλευρά δηλαδή υπάρχει αύξηση της ε, παροχής, αλλά από την άλλη πλευρά διάφοροι φορείς, τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, ε, σε όλα τα επίπεδα, κάνουν προσπάθειες ώστε να μειωθεί η κατανάλωση και για να γίνει αυτό παίρνουν από τον ίδιο πόρο. Ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι δύο αντίθετες ε, τάσεις, ε, χρειάζεται πολύ καλύτερος προγραμματισμός. Τώρα φυσικά εγώ δεν ε, θέλω να σας περιγράψω ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ιδιαίτερα ζωφερό, όχι. Αλλά χρειάζεται να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι οι επενδύσεις που έγιναν, έγιναν σωστά και προσκρούμε στο γεγονός ότι ίσως δεν φτάσαμε στα, επιθυμητά αποτελέσματα γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα σύνδεσης ή υποδομών. Δηλαδή, αν ε, θέλαμε ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αγοράσαμε ένα αυτοκίνητο αλλά δεν ξεχάσαμε να πάρουμε το κλειδί και άρα τα αφήνουμε στο γκαράζ. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο προγραμματισμό θα πρέπει να γίνεται με πολύ πιο ακριβή τρόπο σε σχέση με το παρελθόν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, το συντονισμό ανάμεσα στα κατημέλη, περιφερειακές αρχές, ε, τοπικές αρχές, ε, οικονομικού φορεί. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα σε όλου του ενδιαφερόμενους και μεγαλύτερη συμμετοχή στη φάση του προγραμματισμού. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι. Έτσι θα ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη εισήγηση. Να πω ακόμα μια φορά ποιο είναι το μήνυμά μου. Να μιλήσουμε δηλαδή για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχει προβλέψει 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε συστάσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος, θέλει, επιθυμεί παρακαλώ το λόγο. Για Λασέντα Χατζημαρκάκης. Άλλος παρακαλώ. Προτείνω να λάβουν πρώτα το λόγο αυτοί οι δύο συνάδελφοι και μετά βεβαίως μπορεί να τοποθετηθεί η Κομισιόν. Μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα ε, που την αφορούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Τόιτσα ε, για τις ε, προτάσεις που υπέβαλε που κατά την άποψή μου είναι πολύ λογικές και γενικότερα η έκθεσή του νομίζω ότι κατέστησε σαφές ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς ακριβώς ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, κυρίως ε, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικής ε, Ανάπτυξης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, κυρίως τα νοτιότερα κράτη-μέλη, να έχουν επάρκεια πόσιμου ε, νερού, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αυτό τον τομέα. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν πάνω απ' όλα είναι όπως είπαμε το πόσιμο είδωρ. Όσον αφορά τώρα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, για να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, να τα αποκομίσουμε, θα ήθελα να διατυπώσω μία ερώτηση. Ε, τέσσερις χώρες επελέγησαν, ε, μεσογειακές, πρόκειται για χώρες ε, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής για να προσαρμόσουν ε, την ποιότητα του νερού στις ε, προδιαγραφές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την περίοδο 2002-2006. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία έχουν σχέση με την κατάσταση κατανάλωση αφορούν το έτος 2008. Ήταν η χρονιά ε, κατά την οποία η Ευρώπη, κυρίως οι μεσογειακές χώρες, ε, αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Επρόκειτο ε, για μια έκτακτη κατάσταση. Και θέλω να του ελήφθη το στοιχείο αυτό υπόψη, γιατί χώρες όπως είναι η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, κατά την περίοδο 2007 προσέλκυσε 2 εκατομμύρια μετανάστες, υπήρξε ε, μεγάλη προσέλευση τουριστών. Υπήρχαν λοιπόν ιδιαίτερες συνθήκες, <clears throat> εποχικές αν θέλετε, και βεβαίως ε, στο τέλος του 2007 κανείς δεν περίμενε ότι θα ε, πρόκειται μια τόσο οξία κρίση. Όπως είπε λοιπόν ο συνάδελφος κύριος Τότς, αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καταλήξουμε σε σωστά στοιχεία και να μην ε, στρεβλώνεται η πραγματικότητα. Επίσης, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και συγχαίρω το ελεγκτικό συνέδριο γιατί μπόρεσε να εντοπίσει τόσο την καλή χρήση όσο και ε, παράδοξες εξελίξεις. Ε, είναι σημαντικό ε, να υπάρχει μια καλή πρακτική ε, και αν υπάρχουν οι μετρητές ε, στα σπίτια αυτό επιτρέπει και εξοικονόμηση νερού. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η πρόταση η οποία αφορά στον εντοπισμό υδάτινων πόρων που είναι πιο κοντά στη σταστικά κέντρα, πιο κοντά ε, στο σημείο κατανάλωσής τους. Επίσης είναι καθοριστική σημασία το ε, ελεγκτικό συνέδριο να επιμείνει και εδώ θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν το συνέδριο λοιπόν ε, να επιμείνει στο να κλείσουν οι διαρροές ύδατος. Να, το θέμα των υποδομών είναι καθοριστική σημασίας για να μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα πόσιμου νερού στους ε, καταναλωτές, στους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο ε, Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Ντότσο για την έκθεσή του και κυρίω για το ότι προέβαλε το πόσο σημαντικό είναι το νερό. Είναι πολύ καλό το γεγονό ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, κατάρτισε μια ιδιαίτερη έκτακτη, μη προβλεπόμενη έκθεση για ένα πρόβλημα, όπου όμω θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Και γι' αυτό ζήτησε το λόγο, γιατί αν δει κανεί την έκθεση αυτή, ε, δεν μπορεί κανείς ε, να καταλάβει τι ακριβώς ε, κάνουν τα κράτη-μέλη και τι κάνει η Κομισιόν. Ποιος είναι ο στόχος. Βεβαίως και ε, είναι λίγοι και φιντολοί οι πόροι, αλλά κάποιος στόχος πρέπει να υπάρχει. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους συναδέλφους να ρίξουν μια ματιά στις ενδιάμεσες επικεφαλίδες, που είναι σαφείς. Παραδείγματος χάρη, σελίδα 21 αναφέρεται αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης προς την Κομισιόν. Αυτό δεν συνέβαλε ιδιαίτερα ε, συνέβαλε μόνο σε κάποιο βαθμό. Επίσης λέει στην έκθεση ότι ορισμένες ε, Ορισμένα προγράμματα, επειδή έλειπαν κάποια στοιχεία, δεν εφαρμόστηκαν. Επίσης, αναφέρεται πιο κάτω, ε, σε κάποια προγράμματα υπήρχαν εγγενείς περιορισμοί, άρα δεν λειτουργήσαν τα προγράμματα αυτά. Σε 27 αναφέρεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και αυτό συνεχίζεται. Σε 28 η αρχή της εξοικονόμησης επηρεάζεται από την υπέρβαση κόστους. Σελίδα 29. Ε, περιορίζεται η λειτουργική, το λειτουργικό οικονομικό στοιχείο ενός προγράμματος και το καθεξής. Άρα δηλαδή σε αυτό τον τόσο περιορισμένο τομέα η έκθεση αυτή βρήθη παρατηρήσεων που καταδεικνύουν ότι δεν αντιμετωπίστηκε σωστά το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο εμείς επιτέλους ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιληφθούμε του συνόλου του προβλήματος. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν σε αυτή τη φάση όπου έχουμε νέους επιτρόπους γιατί εδώ ε, ιδιαίτερα αρμόδιο, είναι ο κύριος Χάν, ο οποίο όμως ε, όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα δεν είχε καν να λάβει τα καθήκοντά του. Τώρα λοιπόν πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να πούμε στην Κομισιόν δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα τον αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια πρώτον ότι ε, έγινε πολύ χαλαρή ε, μάλιστα ε, σπάταλη αν θέλετε διαχείριση των χρημάτων αυτό είναι προφανές ε, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κομισιόν πρέπει να αλλάξει πορεία και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να χρησιμοποιούν κονδύλια για προγράμματα τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει κατά τις, μέσα στις επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Ντότζ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι ο κύριο Βόν θέλει το λόγο. Αν είναι κάποιο άλλο συνάδελφο. Όχι, καλώς. Λοιπόν, να σε ακούσουμε εσά μετά την Επιτροπή και βέβαια και το συγκεκριμένο. κύριε Βόν. Πολύ, πρόεδρε, πολύ σύντομα, Πρόεδρε, διότι συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριο εισηγητής που έκανε μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή εκθέση και διεξουδική. Επίση, συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ένα μόνο σημείο πρέπει να πω ότι έχω κάποιες ανησυχίες Ω προ το κόστο του ύδατο. ότι θα πρέπει δηλαδή να επιβαρύνεται με ολόκληρο το κόστος της συντροδότηση ο καταναλωτή, ο πολίτη. Δεν αναλογίζεται το ελεγκτικό συνέδριο τη κοινωνική επιπτώσει ενό τέτοιου μέτρου. Ε, κάποιες οι οποίε ε, μπορεί να είναι φτωχέ, αλλά έχουν πολλά παιδιά και έτσι καταναλώνουν πολύ νερό. Ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη, ε, πάσουν από κάποια νόσο που χρειάζεται να καταναλώνουν πολύ νερό. Δεν θα έπρεπε σε αυτού να δοθεί κάποια διευκόλυνση. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρο. Και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι στις συστάσεις ε, υπαριθμών 1 και 2 και 3 έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένα ε, συγκεκριμένες προτάσεις ή ε, αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ε, και ο συνάδελφος κ. Ντόις έχει κάνει τις προτάσεις από την Επιτροπή. Ποιος θα λάβει το λόγο, κ. Βόλς, κ. Φίστερ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου καταλήγει στο ότι τα διεθνωτικά μέτρα έχουν συμβάλει στη βελτίωση της παροχής ύδατος ε, στα νοικοκυριά με τον ε, διατηθέμενο όγκο, την κάλυψη των δικτύων, την καλύτερη ποιότητα και συνέχεια στην παροχή και την παροχή υπηρεσιών επικεντρώνεται μόνο στα τέσσερα μελη Επιτροπή, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία, που ήταν οι κύριε χώρε ε, που έλαβαν χρηματοδότηση για, τις για την περίοδο αυτή με 29 σχέδια, που αντιστοιχούν στο 13% των συνολικών επενδύσεων ε, ω προ την παροχή υδροδότηση στα τέσσερα ε, εν λόγω κράτη-μέλη. Όσον αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταγραφεί ότι τα κράτη-μέλη έχουν την κύρια και πρωταρχική ε, ευθύνη για την επιλογή και χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων μαζί με τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Διευθυντικού Ταμείου έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πλαίσιο, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο μας στο οποίο κινείται για το το 2007 2007-2013 μόνο παρακολουθεί την ε, διάθεση και λειτουργία των σχεδίων ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές τους. λοιπόν, αν δεν υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές δεν ε, εξασφαλίζεται και αυτό. Το ελέγχουμε με τους ε, καταλόγους που έχουμε προσδιορίσει, καταλόγους δηλαδή επαλήθευσης στοιχείων, την ε, αρχή της ανάκτησης της ε, επένδυσης και με βάση την οδηγία για την διαχείριση των υδάτινων πορών, ιδιαίτερα το άρθρο 9, που είναι υποχρεωτικό από 1η Ιανουαρίου του 2011 για όλα τα κράτη-μέλη. Βάσει αυτής μπορούμε να έχουμε καλύτερη ε, τιμολόγηση της συντροδότησης με βάση την ανάκτηση του κόστους το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής ορυπέρων πληρώνει αλλά και της αρχής της ανάπτυξης κόστους. Ως προς τη λειτουργία των υποδομών που κατασκευάστηκαν με κοινοτική χρηματοδότηση, υπογραμμίζεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν την κυρία, την κυρία ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των σχεδίων και την τήρηση των προδιαγραφών. Ταυτόχρονα όμως και εμείς από πλευράς μας ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι περίπλοκα αυτά τα σχέδια υποδομών και έτσι υπάρχουν ε, κάποιες καθυστερήσεις ενδεχομένω ως προς την παροχή των απαραίτητων στοιχείων, διάθεση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Ως προς τις στάσεις του εισηγητού θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε, και επίσης να δώσουμε κάποιες ε, απαντήσεις στις παρατηρήσεις των βουλευτών. Η οδηγία πλαίσιο για τα είδωρο θεσπίστηκε το 2007 και θεσπίζει ένα πλαίσιο προστασία για όλου του συντάτινου σπόρου, δηλαδή ποτάμια, λίμνες, υδροφόρο ορίζοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να φτάσουμε στο στο επίπεδο του 2015. Η οδηγία προσδιορίζει συγκεκριμένου στόχου ε, τιμών για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2010 καλούνται τα κράτη-μέλη να προσφέρουν συγκεκριμένε προτάσεις ε, με τα σχέδια αυτά λοιπόν, τα οποία αξιολογεί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που εντάσσει συνέχεια στο ε, Γενικό Πρόγραμμα 2012 ε, και την αναθεώρηση για την βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων, βιοπικιλότητα και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υπογραμμίζουμε ότι για το 2013 έχει προσδιορίσει εσωτερική επανεκτίμηση ε, εσωτερικών σχεδίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσφέρει δε τεχνική στήριξη στα κράτη-μέλη, στα νέα κυρίω κράτη-μέλη, όταν ε, προετοιμάζονται αυτά για την υποβολή σχεδίων προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζει τι συστάσει του σημείου 4 του σχεδίου εκθέσεω και υπογραμμίζει ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να προβάλλουν τι ε, εγγυήσει τήρηση του νομοθετικού πλαισίου. Βεβαίως αναγνωρίζετε ότι είναι περίπλοκα τα σχέδια των υποδομών, έχουν πολλές φάσεις και η υποδομή ε, η απαραίτητη υποδομή ίσως να μην εξασφαλιστεί ταυτόχρονα σε κάθε επίπεδο. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθερίσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν. Φυσικά όλα τα σχετικά σχέδια έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην υπόθεση αυτή και υπογραμμίζουμε ότι στην περίοδο 2000-2006 για, ε, με ένα αίτημα μάλλον το οποίο διατυπώθηκε κατόπιν της περίοδου αυτής ε, για την πιο αποδοτική διαχείριση των υδάτων έχει προχωρήσει με μια πρόταση του 2007 στον εντοπισμό και την υλοποίηση μέτρων αποτροπής ε, σπατάλης, δηλαδή απώλειας υδάτων από το δίκτυο, εξοικονόμησης κτλ. Όπως άλλωστε προβάλλονται ως αιτήματα μέσα στο θέμα που μας απασχολεί. Και για να φτάσω στο τελευταίο σημείο, η Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή, σκοπεύει να υιοθετήσει μια ανακοίνωση για την περιφερειακή ολοκλήρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη με στόχο την υπογράμμιση της σημασία των διαφορετικών ταμείων για την παροχή υδροδότηση σε ποσό 8 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 2008-2013 για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήση των υδάτων και τον προσδορισμό προτεραιοτήτων ιεραρχίας αν θέλετε, δηλαδή μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μας ενημερώσατε για την υιοθέτηση της ε, ανακοίνωσης την Δετάρτη μεθαύριο. Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος με τους συναδέλφου, θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς ε, την πρόταση αυτή. Κύριε Βάρη τώρα εσείς, θα σας παρακαλέσω να αντιδράσετε εν συντομία στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις των συναδέλφων, κυρίως τη κυρία Αγιαλά Σέντερ και του κυρίου Βόν και θα σας παρακαλέσω να καταλήξετε στα συμπερασμάτά σα. Κύριε Βάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις της κυρίας Γιώλα Σέντερς, ε, θα ήθελα καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Δηλαδή, το ελεγκτικό συνέδριο ε, ασχολείται με τεχνικά θέματα και αντιμετώπισε τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε ότι έχουμε εξετάσει όλα τα θέματα και έχουμε συζητήσει με εκπροσώπους ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ε, δημόσιων αρχών για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς γίνεται η διαχείριση ε, των υποδομών στα προγράμματα που επιλέξαμε. Το ελεγκτικό συνέδριο πέρα από αυτό χρησιμοποίησε και εμπειρογνώμονες που είναι ειδικοί για τον εφοδιασμό με νερό. Και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Διότι η κυρία Γιάννα Σέντερ, βέβαια και αυτά που είπε είναι πολύ σημαντικά, αλλά όμως κατ' ουσίαν αυτά τα οποία αμφισβήτησε είναι πολιτικής φύσεως θέματα και δεν νομίζω ότι μπορεί να μειώσει κατά κάποιον τρόπο τα στοιχεία που προσφέρουμε εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς ε, ή εσείς αν θέλετε μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα από πολιτική σκοπιά. Αυτό όμως δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αυτό είναι θέμα του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θα εξηγήσει το πολιτικό στοιχείο. Και επίσης θέλω να προσθέσω ότι οι αξιολογήσει του ελεγκτικού συνεδρίου αν δείτε λιγάκι τους πίνακες αφορούν στην κατάσταση πριν από την κρίση και ε, αυτό είναι ένα δομικό στοιχείο. Κατόπιν, όσον αφορά σε αυτά που είπε ο κύριος Βάγκαν, ο οποίος πολύ σωστά επισήμανε το πρόβλημα της ε, κοινωνικής, των κοινωνικών προεκτάσεων αν αυξηθεί το κόστος ε, του νερού. Και όσον αφορά το κόστος αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τη σύνθεση των οικογενειών. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν αγνοεί το θέμα αυτό, γιατί αν δείτε την παράγραφο 68 της έκθεσης, εκεί αναφέρεται το εξή και παραθέτω. Η αρχή της μετακύληση του κόστου στου χρήστε, αυτή είναι μια αρχή η οποία ήταν ήδη γνωστή και εδώ απαντώ και στην Κομισιόν όσον αφορά στο θέμα αυτό. Γιατί η αρχή αυτή προϋπήρχε της θέσης σε ισχύ της οδηγίας πλαίσιο. Και υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο το οποίο παραθέτει η Επιτροπή ε, στο σημείο με 35 όπου Φαίνεται, όπως σας είπα, ότι αυτή η αρχή προϋπήρχε. Όσον αφορά λοιπόν τη μετακύληση του κόστους ε, του νερού στους χρήστες, το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτήν τη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρει ότι ο υπολογισμός του κόστους μπορεί να γίνει έχοντας κατά νου και διάφορους άλλους ε, παράγοντες όπως ε, παραδείγματος ε, χάρη ε, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, αλλά και γεωγραφικά στοιχεία, γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες. Καταρχήν λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι οι κοινωνικές προεκτάσεις. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να μετακυλιστεί το 100% του κόστου στους χρήστες. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην οδηγία πλαίσιο για το νερό του 2004, οδηγία του 2004, Με αυτά λοιπόν νομίζω ότι απάντησα και στις ε, παρατηρήσεις Κομισιόν σχετικά με τη θέση οδηγία σε εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο. Και εμείς πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αυτή η οδηγία ετέθησε εφαρμογή του 2010. Αυτό όμως σας είπα, η αρχή της ανάκτησης του κόστους ήδη προϋπήρχε πριν από τη θέση ισχύ αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γιάννα Θέλετε ακόμη να απαντήσετε, να επανέλθετε μάλλον πολύ στο μα. Ναι, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Θα ήθελα να αντιδράσω, διότι... Γιατί δεν ήθελα να θίξω το ζήτημα τώρα, αφού δεν είχα στοιχεία από το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά μια και το ανέφεραν τώρα, βλέπω ότι στον πίνακα αριθμών 2 έχουμε μια εκτίμηση των καταναλώσεων ε, ε, της κατανάλωσης ύδατος για το 2008 και όπως είπε ο εκπρόσωπος ε, στα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου που απορρέουν από αυτήν την αξιολόγηση στην διάρκεια αυτών των ετών διαπιστώνεται κακή εσφαλμένη αξιολόγηση ως προς τις προβλέψεις του 2008. Για το 2008 λοιπόν Όταν δηλαδή το 2002 έχει ξεκινήσει, ξεκινάει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ε, ε, εμφανίζεται ταυτόχρονα και ένα ποσοστό ανάπτυξης, ε, το οποίο έχει να κάνει και βέβαια με τον τουρισμό. Αύξηση λοιπόν σταθερή και άρα εάν κάνουμε, αν έχουμε να κάνουμε με εκτιμήσεις για το 2008 και από την άλλη ε, συγκρίνουμε αυτές τις εκτιμήσεις ή τις προβλέψεις με την πραγματική κατανάλωση του 2008, καταλήγουμε στο εξή συμπέρασμα, ότι ήταν εσφαλμένες οι προβλέψεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο ή ο εισηγητής λαμβάνουν υπόψη ένα, μια τάση αυξητική στην οικονομία μια ανάπτυξη ως πρόβλεψη ενώ τελικά το 2008 εμφανίζεται κρίση οικονομική και πώς προσαρμόζει αυτές τις προβλέψεις στο ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω πόσο τεχνικό είναι αυτό το ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είμαστε θέση να προβούμε σε μια πολιτική αξιολόγηση. Άρα πρέπει ή μη τι άλλο σε τεχνικό επίπεδο να γνωρίζουμε εάν οι προβλέψεις και η πραγματική κατανάλωση που καταγράφεται εκ των υστέρων είναι ορθές ή όχι. Ή θα έπρεπε να συγκρίνουμε μια κάποια περίοδο που βρίσκεται εκτός οικονομικής κρίσεως. Ο Πρόεδρος. Ναι, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο ασφαλώ θα μας απασχολήσει και στο έγγραφο τη απαλλαγή. Ο κύριος Δόιτς ε, πρόσεχε βέβαια με παρακολούθησε με πολύ προσοχή τα όσα υπόθηκαν και Δόιτς παρακαλώ για να καταλήξουμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κλείσω με τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις εξαίρετες ε, προτάσεις τους. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παρόντες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εντατική η συζήτηση. Βλέπω με ικανοποίηση ότι συμφωνούμε εδώ στην Επιτροπή μας ότι ε, είναι ε, ως προς την προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε για τα υδάτινα αποθέματα. Δηλαδή συμφωνούμε ότι στον 21ο αιώνα το είδωρ είναι στρατηγική σημασίας πόρος και γι' αυτό ε, απαιτείται να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτο η διαπίστωση αυτή. Δεύτερη, ε, η κυρία Γιάλα Σέντερ έθεσε ένα άλλο ζήτημα, ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία και δεδομένα. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, όπως άλλωστε και εγώ, υπογράμμισε αυτό το στοιχείο. Χρειαζόμαστε εκτιμήσεις στέρεες, σωστές, για να έχουμε ε, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην δουλειά μας. Άρα χρειαζόμαστε καλύτερες εκτιμήσεις. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Τρίτον, άκουσα τα όσα είπε ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω έθιξε την ίδια ιδέα και ο κ. Χατζημαρκάκης Καταλήγουμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα σαφές σύστημα ελέγχου και μια και μιλούμε για έναν στρατηγική σημασία φυσικό πόρο και με δεδομένο ότι οι υποδομές ε, της υδροδότησης φτάνουν στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να σας το δώσω παραστατικά, έχουμε να κάνουμε με τη βιτρίνα της δουλειάς που κάνουμε. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα αγαθό το οποίο φτάνει στον κάθε πολίτη και που καθιστά ορατό το τι κάνουμε για τον κάθε πολίτη. Άρα χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλούς ελέγχους, ορατούς ελέγχους, διαφανείς ελέγχους προς την χρήση των πόρων και εν τέλει, όπω ανέφερε ο κύριο Βόν, θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερε πληροφορίε σε λεπτομέρειε για τα όσα έθιξε εκείνο, κυρίω όσον αφορά την τιμολόγηση του ύδατο. Ναι, αυτά που λέει το Ελεκτικό Συνέδριο βεβαίω είναι προφανή και λογικά πιστεύω κατά την άποψή του, ότι δηλαδή είναι χαμηλέ οι τιμέ. Πλην όμω, ο κύριο συνάδελφο ανέφερε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι δηλαδή η παροχή υδροδότησης και χωρίς να πρέπει να κρίνουμε αν είναι καλή ή κακή η πορεία που σημειώνεται στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή η πορεία της ιδιωτικοποίησης, ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές. Ότι ο Ριπένον πληρώνει, ότι επιβάλλεται η αρχή της περιβαλλοντικής προστασίας, ότι έχουμε να κάνουμε με αγαθό δημόσιο, στο οποίο έχει δικαίωμα ο πληρωνει οτι επιβαλλεται η ένας, καθαρό δηλαδή, πόσιμο νερό Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζονται και δεν μπορεί μια οικογένεια πιο φτωχή από τι άλλε να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Δεν μπορεί να υποφέρει μια οικογένεια μόνο και μόνο λόγω τη οικονομική επιφάνεια. Εάν δούμε λοιπόν από την άλλη πλευρά στην ε, δεδομένη την ιδιωτικοποίηση, την ιδιωτική εταιρεία η οποία θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδο τη, έχουμε να κάνουμε μια πολύ λεπτή ισορροπία την οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προκειμένου να δώσουμε τις βασικές αρχές που θα ισχύουν για το ε, σύστημα παροχής αυτής της υπηρεσίας. Αυτές οι βασικές αρχές δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Νομίζω ότι υπογραμμίζει αυτό και, η αρχή των, και το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και η δική μου έκθεση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ε, κλείσουμε το θέμα αυτό προσωρινά. Αν και ίσως ο κύριος Βάρη θέλει πάλι το λόγο. Όχι. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα στην έννοια της ημερησίας διάταξης και ε, περνάμε αμέσω στο σημείο υπαριθμών 6 και θα ρωτήσω την κυρία Ματσιού και την κυρία Κιώστιγκερ εάν συμφωνούν για το κατοπροσδιορισμό τη ημερησία διάταξη για τις Συνεδρίες Οι σοσιαλιστέ δημοκράτες ζήτησαν πρώτα να συστηθεί το σημείο 6 και μετά το σημείο πέντε πρώτα, εκ τη κυρία Ματσιού και μετά τη κυρία Κρέστινγκερ. Αν δεν έχετε τη κυρία Ματσιού, να κάνουμε την αντιστροφή στην ημερήσια διάταξη, αλλά βλέπω ότι ε, συνενείται και οι δύο. Α περάσουμε λοιπόν στο σημείο 6. Δηλαδή το θέμα της ε, παρακολούθησης της άρνησης απαλλαγής για την ε, Αστυνομική Ακαδημία, για την περίοδο 2008. Πρόκειται για ένα ε, έργο με πολλές πράξεις κυρία Ματσιό έτσι δεν είναι έχουμε να κάνουμε με μια άρνηση απαλλαγής, έχουν ακολουθήσει πολλές συζητήσεις. Σε επίπεδο συντονιστών είχαμε συμφωνήσει ότι θα χρειαστεί ασφαλώς μια νέα έκθεση και με παρουσία των εκπροσώπων του Λεπτικού Συνεδρίου αλλά και των διευθυντικών στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας θα πρέπει να γίνει συζήτηση για την προετοιμασία του πεδίου και παρακαλώ τώρα την κυρία Ματσίρα λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η τέταρτη ακρόαση σε επίπεδο Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, γιατί έγινε και στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ε, κατόπιν αιτήματο του κ. Μπισούτη, λέει, ε, ακρόαση, ύστερα από την ε, γνωμοδότηση για την απαλλαγή 2009 Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει κάρτα περιορίστων διαδρομών ο διευθυντή τη ε, Αστυνομική Ακαδημία, αφού θα έρχεται τόσο τακτικά σε εμά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, 30 Νοεμβρίου είχαμε αυτή την ακρόαση, που όμω δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε το Governing Board, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ήμασταν τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και μάλιστα, ο πρόεδρο ήθελε να επαναληφθεί αυτή η ακρόαση. Εν πάση περιπτώσει, όσο με αφορά, ο κύριο Μπομφή, ο διευθυντή, ε, εντωμεταξύ μας έδωσε τι απαντήσει στα ερωτήματά μα. Εγώ δεν έχω πλέον απορίε προ ε, τον ε, διευθυντή τη Αστυνομική Ακαδημίας. Θα ήθελα όμω να ακούσω τον πρόεδρο του Governing Board, του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κύριο Μαρίνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του οποίου τη φωνή δεν έχουμε ακούσει ακόμη και πιστεύω θα φωτίσει με τι απόψει του, ε, του συναδέλφου. Δεδομένου ότι ο κύριος Μαρίνη συνεδριάζει, συμμετέχει σε αυτό το governing board. Ο κύριος Μποντάν δεν είναι ο ε, εκλεγής πρόεδρος αυτού του governing board. Μόλις ανέλαβε καθήκοντα του νέου governing board καλύτερα και να σα το ένα πολύ στομό ε, ιστορικό της υπόθεσης, αγαπητοί συνάδελφοι, με την Αστυνομική Ακαδημία είχαμε το εξής το 2007 επί Πορτογαλικής Προεδρίας λαμβάνει η Πορτογαλική Προεδρία ένα ανώνυμο ε, γράμμα, μια ανώνυμη επιστολή, την οποία αποστέλει και στην ε, Όλαφ και στην ε, Τριανδρία, στην Τριμερή, ως προς κατηγορίες, περιλαμβάνει αυτή η επιστολή, για κακοδιαχείριση στην αστυνομική Ακαδημία. Και καλείται να αποσταλεί αυτή η επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πριν από τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρία, ο πρόεδρος διατυπώνει ένα σχέδιο δράσης και παρακολούθησης της υπόθεσης. Ε, παρουσιάζεται από την Επιτροπή μια έκθεση πεπραγμένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας ενημερωνόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από την GLS των ευθυνών της ε, η αστυνομική, ακαδημία μάλλον καλείται να διευ κρινήσει και να επιλύσει τα εσωτερικά τη προβλήματα. Δεν γίνεται τίποτε τέτοιο και η Τσεχική Προεδρία αποστέλει στην νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή όπου ζητεί αρρωγή και επίσημη τοποθέτηση, γνωμάτευση δηλαδή. Και στη συνέχεια το 2010 αποστέλλεται ε, μνημόνιο με τι ε, καταγγελίε ει βάρο του Διευθυντή και την αδυναμία συνεργασία σε συνθήκε απορρίτου και εμπιστευτικότητα με τον κύριο αυτόν. Η Σουηδική ε, Προεδρία αντικαθιστά ε, τον Διευθυντή ε, και ζητεί την παρέμβαση της ΟΛΑΦ και τη συνέχεια τη γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Ποτέ, εσείς ήσασταν παρόν το 2006, 7 και 8 ήδη, ε, ύστερα από τα όσα είδαμε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Καθολοσορίζω εδώ και τον κύριο Φιέλερ που ήρθε και είχε την εισήγηση το 2007 στην υπόθεση αυτή. Θα μπορούσατε νομίζω να μας διαφωτίσετε ίσως κύριε Μποντάνη για το πώς εργάζεται αυτό το Governing Board, διότι έχουν διατυπωθεί πολλές καταγγελίες για τον τρόπο δράσης του προηγούμενου διευθυντή, αλλά εμένα με ανησυχεί και ο τρόπο εργασία του ίδιου του Governing Board. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά αυτά που μαθαίνουμε και νομίζω ότι υπήρξε μια κάποια ελαφρότητα χειρισμών. Και μόνο η Σλοβενική Προεδρία με την ε, αντίδρασή τη και την ανώνυμη επιστολή που προκάλεσε αυτή τη σειρά αντιδράσεων με την ε, τσεχική προεδρία μας οδήγησαν τελικά σε αυτές τις εξελίξεις, διότι έχουμε και αμέλεια και κακοδιαχείριση οικονομική, για να μην μιλήσω για υπεξαιρέσει από πλευράς του ε, πρώην διευθυντή, αλλά έχουμε και ζήτημα μη εκτέλεσης του έργου που έπρεπε να έχει εκτελέσει ο προηγούμενο διευθυντή. Επίσης έχουμε ζήτημα κακού συντονισμού μεταξύ των μελών του Governing Board ε, απουσία σοβαρότητα στη δουλειά αυτήν. Η δε Γαλλική Προεδρία η οποία διακήρυσε τεκμήριο αθότητας προσπαθώντας να αποφύγει μια τοποθέτηση στην εποχή εκείνη νομίζω μας ε, υποχρεώνει να πούμε ότι ναι βεβαίως πριν να ε, κατηγορηθεί, μάλλον πριν να καταδικαστεί ο οσδήποτε θεωρείται ότι είναι αθώος και ισχύει το τεκμήριο αθότητας αλλά δεν μπορούμε και να παραβλέψουμε τα όσα έχουν συμβεί σε αυτή την υπηρεσία. Και λυπούμε διότι ο προκατοχό σα δεν μας ενημέρωσε καθόλου σε όσα ζητήματα είχαμε ζητήσει πληροφορίε. Εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματσιέ. Πολύ συγκεκριμένες άμεσες ερωτήσεις και απευθύνονται βεβαίως σε εκπροσώπους της Αστυνομική Ακαδημίας, της ΕΠΟΛ. Πριν ακούσουμε τον κύριο Μποντεά και τον κύριο Μπονφι παρακαλώ και το ελεγκτικό συνέδριο η κυρία στον κύριο Ορσίαν έχει ε, κάτι να προσθέσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα την άδειά σας ε, να ακούσουμε τον ε, κύριο Ποφούμ και τους συναδέλφους του από την ΣΕΠΟΛ. Τι θέλετε, κύριε Μπράιν Γκρέι, να ακούσετε πρώτα τις απαντήσεις. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Ας δώσουμε το λόγο σε εκείνους στους οποίους απευθύνθηκαν οι ερωτήσεις. Εκπροσώπος του ΣΕΠΟΛ, κύριος Μποντέ, που είναι εκπρόσωπος του Δικαιωτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε όλοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής Καταρχήν να σας πω ότι είναι τιμή μου που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για τα βήματα στα οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε βήματα ώστε να διορθώσει τα σφάλματα που έγιναν στο παρελθόν. Τα ακούσατε να παριθμώνται από την εισηγήτρια. Θα ήθελα δε να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της ΣΕΠΟΛ, διότι ε, καταναλώνει τόσο πολύ χρόνο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει, έπρεπε τόσο πολύ να σας απασχολούμε. Επειδή είμαστε αστυνομικοί, θα πιστεύω ότι θα έπρεπε εμείς πρώτοι από να συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία. Τώρα, ε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία δημιουργήθηκε το 2001 και αρχικά χρηματοδοτείται από τους προπολογισμούς των κρατών μελών. Στην Κοπεχάγη το 2001 ε, η γραμματεία δεν ήταν μόνιμη και ο πρώτος προϋπολογισμός για την ΣΕΠΟΛ φτιάχτηκε το 2002 από 15 κράτη-μέλη. Το 2010 ε, προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 νέα κράτη-μέλη και άρα ο προπολογισμό μας αυξήθηκε σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και με βάση η απόφαση του Συμβουλίου, η ΣΕΠΟΛ χρειάστηκε να φτιάξει μια μόνιμη γραμματεία με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει εκεί και έχετε επισκεφθεί την ε, γραμματεία της ΕΠΟΛ. Βρίσκεται στη μέση του ποθενά, αυτό το κτίριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να μεταβεί στο συγκεκριμένο μέρος. Δεν, έχουν, δεν υπάρχουν συνδέσεις, δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επικοινωνία, δηλαδή ο κόσμος που εργάζεται εκεί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, στα τέλη του 2005 η γραμματεία της ΕΠΟΛ είχε φτιαχτεί, είχε καταρτιστεί με 15 μόνιμους υπαλλήλους και ξεκίνησε να εργάζεται. Τότε ο προπολογισμό ήταν 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Ε, τώρα, μετά από το 2006 γίναμε οργανισμός, ευρωπαϊκός οργανισμός με απόφαση του Συμβουλίου και τότε κιόλα ο προϋπολογισμός μας αναλύθηκε, ε, αξιολογήθηκε από την ε, Κομισιόν και καθώς και η απορρόφηση αυτού. Τότε το Δικητικό Συμβούλιο θεώρησε πως ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή, ο έλεγχος δηλαδή των λογαριασμών μας. Ε, είχαμε λοιπόν προβλήματα μέχρι το 2007, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τη γραμματεία και με τον διευθυντή. Ορισμένα μέλη ξέφρασαν τις ανησυχίες τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση και αποφάσισε ότι ο διευθυντής έπρεπε να προβεί στα απαραίτητα βήματα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Η κυρία Ματιού ανέφερε επίση ότι όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου του 2007, πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που μας παρουσίασε τα προβλήματα. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας διετάχθη ο Διευθυντής από το Διοικητικό Συμβούλιο να διορθώσει την κατάσταση. Το δεύτερο ήμεση του 2008 και αρχές του 2009 έγιναν πολύ αυστηροί έλεγχοι, τους οποίους ε, διέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο διότι αποκαλύφθηκαν σφάλματα και στην Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τη δημοσιονομικά του οργανισμού. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει μια ελεγκτική ομάδα, μια ειδική ελεγκτική ομάδα. Και αυτή η ομάδα θα είχε το έργο του ελέγχου όλων των οικονομικών συναλλαγών του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια δε της τσεχικής προεδρίας Υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση μετά από μια σειρά γεγονότων. Ο διευθυντής χρειάστηκε να παρετηθεί λόγω των, της κακοδιαχείρισης που είχε διαποστοθεί και των σφαλμάτων στα οποία είχε ε, πέσει ο ίδιος. Και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Ιουδικής Προεδρίας υπήρξε μια μεταβατική περίοδος με έναν ε, ε, αναπληρωματικό διευθυντή και στο τέλος του έτους εξελέγει νέος διευθυντής, ο κύριος Μπάνφι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτοτε ο κύριος Μπάνφι είναι ο διευθυντής του οργανισμού, ο οποίος έχει δείξει μεγάλο επαγγελματισμό έχει κερδίσει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μεταμορφώσει τη διαχείριση ε, του ε, ΣΕΠΟΛ και επίσης ε, την, τον δημοσιονομικό έλεγχο προσέλαβε νέους ειδικού για την οικονομική διαχείριση του οργανισμού οι οποίοι προσπάθησαν να διορθώσουν όλα τα σφάλματα. Λειτουργούν δηλαδή αναδρομικά και ό,τι ήταν νομικά ε, δυνατόν προσπαθούν να το διορθώσουν. Ελπίζω λοιπόν πως οι προσπάθειες τις οποίες προέβη η νέα γραμματεία ο νέο διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτιμηθεί. Φυσικά συνεχίζεται η προσπάθεια λόγω όλων αυτών των γεγονότων. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας ακόμα. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλες αυτέ τις υποθέσεις μέσα στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Υπήρξαν θετικές ε, αλλαγές ε, βεβαίως μέσα στην ΣΕΠΟΛ που στη σωστή κατεύθυνση το περασμένο έτος το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες ιδέες που πρότεινε ο Διευθυντής που στόχο έχουν την αναδιάρθρωση της γραμματείας ώστε να λειτουργεί αυτή πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει ένα νέο στατηγικό σχέδιο επίσης που έχει οθετηθεί και έχουμε αναπτύξει και ένα νέο εργαλείο, ένα μέσο παρακολούθησης που στενά παρακολουθεί την εφαρμογή και την υλοποίηση των ε, προγραμμάτων μας. Έχουμε επίσης ε, αναθέσει σε εξωτερικούς ε, συνεργάτες να συντάξουν έκθεση για την πενταετή περίοδο για μια πενταετή περίοδο που θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο και θα αναλύει την περασμένη πενταετία δραστηριότητας της Apple, συν θα περιλαμβάνει προτάσεις για το μέλλον. Με βάση τις συστάσεις που μας έχει υποβάλει η Κομισιόν, το Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Επίση, προγραμματίζουμε από κοινού με την Κομισιόν να κάνουμε τα εξή κατά τη διάρκεια τη Ουγγρική Προεδρία, να διοργανώσουμε μία διάσκεψη που θα εστιάσει στι δραστηριότητε τη ΕΠΟΛ, μια μονοήμερη διάσκεψη, ώστε να συζητήσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημίας. Θέλουμε να προβούμε σε όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Ελπίζω λοιπόν να μπόρεσα έτσι να σας εξηγήσω όλες τις προσπάθειες, το ιστορικό και ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και καθώς και το ποιο μέλλον θα θέλαμε να δούμε όσον αφορά την συνεργασία. Όλα αυτά τα λέω και εξ ονόματος της ε, γραμματείας αλλά και της διοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικό, αλλά νομίζω ότι οι ερωτήσεις κυρίας Ματιό απαντήθηκαν. Βεβαίως, αν θέλει μετά μπορεί να ζητήσει το λόγο, Τώρα όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάνφη, ελπίζοντας ε, ότι θα απαντήσει σε αυτές τις ειδικέ ε, ερωτήσεις κυρίας Ματιό. Μετά, το λόγο έχει στήσει ο κύριος Φιένα, άλλος παρακαλώ. Ε, κύριε Μπάνφη, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως ε, αναφέρθηκε, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι εδώ ε, και μπορώ να σας παρουσιάσω την έκθεση της Αστυνομικής Ακαδημίας ε, σχετικά με την επίτευξη, την πρόοδο του προγραμματός μας. Η αλήθεια είναι, πριν από κάποια χρόνια ονειρευόμουν να έρθω κάποτε στο Κοινοβούλιο και να το δω από κοντά πώς είναι. Τώρα βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει κανείς εδώ μέσα. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να έχω πιο ευχάριστη παραμονή στο Κοινοβούλιο. Αυτά που κληρονόμησα δεν είναι και εύκολα. Βέβαια δεν μπορώ να πω και ότι η αποστολή μου είναι αδύνατη, mission impossible, κάθε άλλο. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και διορθώνονται πάλι από ανθρώπους ενδεχομένως με μεγαλύτερη στράτευση, επαγγελματισμό, πνεύμα συνεργασίας και θέλω να ελπίζω και με κάποια κατανόηση εκ μέρου σας. Κανείς δεν αμφισβητεί ε, το σύστημα εκπαίδευσης το ευρωπαϊκό για την ε, δίωξη του εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει αυτούς τους θεσμούς και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μπορώ και εγώ ε, να συμμετέχω στις ε, αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο αποφάσισε και υποβλήθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί το τρίτο πρόγραμμα δράσης, ε, ένα πρόγραμμα που το είχε ζητήσει το Συμβούλιο, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και ε, κατόπιν συστήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Τότε λοιπόν η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έλεγξε την δεύτερη έκθεση πρόοδου, τη δική μας, και κατέληξε στο ότι η ΣΥΠΟΛ σωστά εφαρμόζει το πολιτες πρόγραμμα και τότε η Αστυνομική Ακαδημία, η ΣΥΠΟΛ, ε, δεν έλαβε αρνητικές παρατηρήσεις. Εξάλλου αναφέρθηκε ότι κάποια σημεία ε, έπρεπε να διευκρινιστούν ε, περαιτέρω. Εγώ συμφώνησα και καταλήξαμε με την Υπηρεσία Ιστορικού Ελέγχου να κάνουμε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε αυτά τα ορόσημα, αν θέλετε, να γίνουν πιο ορατά στο μέλλον. Κατά την τελευταία κρόση που έλαβε χώρα εδώ, ελπίζω να δώσαμε ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις κυρίας Ματιό. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες ε, προσαρμογής ε, λαθών από τα προηγούμενα έτη και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ενημερώσω ότι ο νεοδιορισμένος ε, ορκωτός λογιστής ε, και οι αρμόδιοι του προπολογισμού βρίσκονται εδώ. Αν λοιπόν έχετε κάποιες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να σας δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Ας δούμε τώρα λιγάκι γιατί δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις που υπήρχαν στην Ακαδημία. Μέχρι το τέλος του 2010, το Δεκέμβρη του 2010, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καθυστερήσεις του 8 και του 9. Η ΣΥΠΟΛ είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις ε, τηρώντας τις ε, προθεσμίες ίσως ε, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων να προέκυψαν κάποιες καθυστερήσεις που δεν είναι όμως σημαντικές. Συνεχίσαμε επίσης να δουλεύουμε για την ενίσχυση της γραμματείας. Αν κάποιος ασχολήθηκε ποτέ με το να προσλάβει με βάση τους, ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα έχει καταλήξει ότι χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες για να μπορεί κανείς να επανδρώσει μια υπηρεσία όπως εμείς στη γραμματεία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το 2010 μετά το διορισμό μου προσλάβαμε εννέα προσωρινούς υπαλλήλους επιλέξαμε επτά εθνικούς εμπειρογνώμονες Έχουμε και άλλες οκτώ διαδικασίες πρόσληψης που τρέχουν. Αυτή λοιπόν τη στιγμή από τις 26 ε, θέσεις προσωρινών υπαλλήλων, οι 20 έχουν ήδη καλυφθεί. Επίσης, λάβαμε την ε, τελική έκθεση της Μούρεν Στέφανς που εντρεύει στο Λονδίνο σχετικά με τις ε, ιδιωτικές ιδιωτικούς πόρους. Και εκεί επιβεώνεται αυτό ε, που είπε ο πρώην διευθυντής της ΥΠΟΛ. Βέβαια υπήρχαν κάποιες διαφορές στα στοιχεία, όμως εμείς δεχθήκαμε τα απορίσματα του εξωτερικού ελέγχου. Και επιπλέον ε, ζήτησα από τον πρώην διευθυντή να συμφωνήσει με την ε, νομική θέση που έλεγε, που ανέφερε ότι άτομα που χρησιμοποιούν ταξί για να πάνε στο αεροδρόμιο δεν ήξεραν ότι αυτό ήταν παράνομο και ρυθμίστηκε εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό από πρώην διευθυντές και δεν υπήρξε κανός είδου συνωμοσία. Ε, νόμιζαν ότι παίρνοντα ταξί ε, δεν παραβιάζουν κανένα κανόνα. Όμως ε, βέβαια και κάποιος ε, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη ζημιά που προκλήθηκε. Γι' αυτό και εξέδωσα αυτή την ανακοίνωση. Βέβαια δεν έχει λήξει η προθεσμία και η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Επίσης βελτιώσαμε σημαντικά τις προμήθειες, το θέμα των προμηθειών. Εγώ ενέκρινα ένα εγχειρίδιο προμηθειών το οποίο επεξεργαστήκαμε μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ε, αδελφούς οργανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα τους χαρακτηρίσω. Επίσης, ε, εισαγάγαμε συμφωνία πλαίσιο όπου περιλαμβάνονται θέσεις για εκπαιδευτές που αυτό ήταν τελικά και η πηγή της κριτικής που είχε ασκηθεί κατά τους προγενέστερους ελέγχους. Τα συμβόλαια αυτά ανάμεσα στα μεμονωμένα άτομα και τους εθνικούς φορείς εκπαίδευσης, όχι ανάμεσα σε μεμονωμένα άτομα και τη ΣΥΠΟΛ, αυτές οι συμβάσεις ε, εξέπνευσαν το 2009 και δεν ανώθηκαν. Όσον αφορά τώρα τις ε, εξαιρέσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν εγκρίθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν ε, η διοίκηση τώρα ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο ε, να διαγράψει κάποιες παραγράφους από τον οικονομικό κανονισμό της Ακαδημίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε κάποιες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Πολύ σωστά επισημάνθηκε επανειλημμένα ότι το σύστημα εσωτερικών ελέγχων δεν εφαρμόζεται σωστά. Και κάτι που επιτεύχθηκε πολύ σημαντικό είναι ότι οι αρμόδιοι αυτού του εσωτερικού ελέγχου ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανασυστήθηκε ο εσωτερικός έλεγχος και αυτοί έχουν αναλάβει να να καταθέσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόγραμμα ε, το οποίο ε, θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου το Μάρτιο. Δυστυχώς ε, η επιλογή του υπαλλήλου εσωτερικού ελέγχου δεν ολοκληρώθηκε. Στην αρχή πρόσφερα αυτή τη θέση σε έναν θαυμάσιο υποψήφιο. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος αυτός ε, είχε υποβάλει τα χαρτιά του και στι Βρυξέλλε ε, και έλαβε μια πιο ελκυστική προσφορά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, ξεκινήσουμε από την αρχή όσον αφορά την επιλογή του υπαλλήλου αυτού. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι ο δικός μου στόχος δεν είναι να ισχυριστώ ότι όλα βαίνουν καλώς στη ΣΥΠΟΛ. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Μπορέσαμε να διασφαλίσουμε την ευνομία, μπορέσαμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά δεν είμαστε τέλειοι για μένα και για όλους τους ε, συναντέλφους που εργάστηκαν ιδιαίτερα σκληρά κατά τα περασμένα έτη. Εμείς ήμασταν τα θύματα των λαθών και νομίζω ότι μας αξίζει υπομονή απέναντι στο πρόσωπό μας, όχι βέβαια ανοχή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ε, εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την απαλλαγή και τις προσδοκίες. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα ήταν να ανακτήσω την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι σαφές, γιατί ε, ε εμπιστοσύνη, αν δεν υπάρξει απαλλαγή, δεν μπορούμε να προσφέρουμε ικανοποιητική εκπαίδευση και μάθηση ε, στην ευρωπαϊκή κοινότητα στους αστυνομικούς, ευρωπαίους αστυνομικούς ε, δίωξης εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιέρνερ. Έχετε εσείς το λόγο τώρα. Θα ήθελα Πρόεδρε, να ευχαριστώ καταρχάς και το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ε, Διευθυντή για τα σχόλιά τους. Όταν ε, έχει παρακολουθήσει κανείς την υπόθεση αυτή ε, για ένα διάστημα, είναι περίπου σαν αυτό που είχε τη συνήθεια να λέει η μάνα μου, ότι εξηγήσει πολλές, δικαιολογίες ολίγες. Καταλαβαίνω τις εξηγήσει, ε, το απόκεντρο της τοποθεσίας κτλ. Αλλά, αλλά, δεν υπάρχει πλήρης εξήγηση. Και πάντως δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Γεγονός όμως είναι ότι πρόκειται για μια μικρή αποκεντρωμένη υπηρεσία η οποία έχει αναλάβει μεγάλο κομμάτι ενός δημοσιονομικού κανονισμού. Και παραλαμβάνω δεν αποτελεί αυτό ε, δικαιολογία διότι όπως και να έχει κατάσταση οφείλει να τηρεί τους κανόνες που ισχύουν 100% χωρίς καμιά παρέκκληση. Πλην όμως αυτό που πάλι ε, ακολουθεί σαν συλλογισμό είναι ότι μάλλον έτσι θα είναι πάντα τα πράγματα. Χωρίς να έχω παρακολουθήσει ε, το γίγνεσθε σε άλλε αντίστοιχε μικρές ε, υπηρεσίες, διαιρωτώ με μήπως τελικά το πρόβλημα είναι ε, ζήτημα μεγέθους και αν είναι ζήτημα μεγέθους μήπως αξίζει τον κόπο να καταργηθεί η ΣΕΠΟΛ, η αστυνομική αστυνομία και το έργο της να αναλάβει κάποια άλλη, να συγχωνευτεί ενδεχομένως. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες ευκαιρίες και η Επιτροπή είχε προσφέρει υποστήριξη σε ε, μικρότερες περιφέρειες. Είχαμε συζητήσει σε περίπτωση μιας προηγούμενης απαλλαγής ε, ότι οι μεγαλύτερες περιφέρειες θα μπορούσαν να συγχωνευθούν με μικρότερες υπηρεσίες, αλλά με προϋπόθεση ότι θα επιλύονται και τα πρόβλημα. Εάν δεν επιλύονται, γιατί να γίνει συγχώνευση. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους παρόντες εδώ εκπροσώπους ή συναδέλφους ε, έχει να κάνει αντίστοιχα σχόλια στο θέμα αυτό. Άλλωστε ήταν καλό να κάνουμε μια απογραφή του τι είδους ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες έχουμε. Ευχαριστώ κύριο Γκάια. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω ακριβώς τα όσα είπε ο κύριος ε, Φιέλνας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή καθηκόντων της αστυνομικής ε, ακαδημίας, την οποία ασφαλώς δεν αμφισβητούμε και δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε εδώ. Έχουμε να κάνουμε με ένα εσωτερικό χώρο μέσα στον οποίο η αστυνομία, που πάντα θα είναι εθνική και πρέπει να παραμείνει εθνική, θα έχει ένα κοινό επίπεδο ε, κατάρτισης, επιμόρφωσης για να μπορεί να συνεργάζεται, να συνεργάζονται δηλαδή, τα αστυνομικά στελέχη μεταξύ τους και οι υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουν τις τάσεις ε, και το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να το επιτελέσει κατά καλύτερο τρόπο μια ιδιαίτερη ακαδημία που θα έχει αυτό το καθήκον ή μια υπηρεσία η οποία θα έχει παραδείγματι συγχωνευτεί μέσα στη Europol, είναι μια άλλη ιστορία και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δούμε τα θέματα αυτά. Και γι' αυτό, δεδομένου ότι έχει προεξαγγείλει και μια έκθεση το ελεγκτικό συνέδριο, θεωρώ ότι είναι καλό να συζητήσουμε για άλλη μια φορά το θέμα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, να δούμε τι καθοδήγησε μας το ελεγκτικό συνέδριο και πώς θα πρέπει να, σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είναι βέβαιο ότι όταν έχουμε συνεργατική ε, δράση, ε, κερδίζουμε, ξεκονομούμε από τους πόρους μας, από τα κονδύλια, αλλά εάν κάτι δεν ταιριάζει και δεν μπορεί να ε, λειτουργήσει μαζί με κάποιο άλλο, με κάποιο άλλο τομέα αρμοδιοτήτων, ας μην επιδιώκουμε με το ζόρι συνεργατικές λειτουργίες και συνέργεια. Αυτό. Κατά τα άλλα, ελπίζω να δούμε και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου στοιχεία ουσιαστικά τα οποία θα εμπλουτίσουν τη συζήτησή μας στο, στο θέμα αυτό. Και εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Τώρα, ως προς τις δύο εκθέσεις και τα όσα άκουσα από την Αστυνομική Ακαδημία. Σημειώνω καταρχάς ότι περιμένω να δω και τις αντιδράσεις της Επιτροπής Βλέπω ότι το, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κύριος Μπάνφη δηλώνουν πως είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν ε, χειρισμό και να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακά τα όσα ακούσαμε, το ότι χρειάζεται δηλαδή για να αλλάξει η κατάσταση στην αστυνομική ακαδημία. Δεν έχουμε προχωρήσει πιστεύω τόσο ώστε να διαπιστώσουμε ότι έχουν επιληθεί τα προβλήματα, πλην όμως τουλάχιστον εγώ προσωπικώς μπορώ να αισθάνομαι αισιοδοξία από τα όσα ακούω πλην και από την άλλη ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει αλλάξει η κατάσταση με το 2008 και το 2009 έχοντας υπόψη και άλλωστε το είπατε και σε ένα βαθμό ότι ήσασταν ούτως υπήν θύματα, δηλαδή κληρονομήσατε προβλήματα που έχετε να επιλύσετε τώρα. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε και όταν έρθει η ώρα για την απαλλαγή θα πρέπει να αναγνωριστεί και να κρυθεί αντίστοιχα το χρονικό σημείο μέσα στο οποίο αναλάβατε καθήκοντα. Αλλά αυτή δεν είναι η στιγμή τώρα. Τώρα έχουμε να συζητήσουμε την περίοδο 2008-2009. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από αυτή την περίοδο βεβαίω προχωρούν προ επίλυση, αλλά αυτή την ε, απαλλαγή έχουμε να συζητήσουμε. Και έχω μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε τι συμπεράσματα καταλήγει. Την έχω υποβάλει την ερώτηση και η απάντηση που έλαβα από τον Επίτροπο ήταν μάλλον απογοητευτική. Είμαι νεοεκλεγέν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και διαπιστώνω ότι υπάρχουν δυσκολίε και προβλήματα σχέση με τι αποκεντρωμένε υπηρεσίε. Όταν λοιπόν διατυπώνεται το ερώτημα τι είδου θεσμικά συμπεράσματα διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτά τα προβλήματα, σε τι συμπεράσματα καταλήγει, απάντηση δεν έχω πάρει. Εγώ δεν το δέχομαι όμω αυτό, να μην δίνεται απάντηση, γιατί βεβαίω ναι, ισχύουν οι συνθήκε, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει όταν υπάρχουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες ε, οι οποίες δεν έχουν απορροφή στα χρήματα του, Ευρωπαίου Φορολογούμενου κατά τον δέοντα τρόπο, θα πρέπει να καταλήγει σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τη λειτουργία και την ύπαρξη αυτών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ομολογώ λοιπόν ότι με κατέπληξε πολύ αρνητική επιτροπή. Δεν έδειξε διάθεση να καταλήξει τέτοιου συμπεράσματα και μέτρα. Και θα ήθελα και εδώ παρόντες εκπρόσωποι της Επιτροπής να ε, μας εξηγήσουν πώς αναπτύσσεται ο εσωτερικό διάλογος για το θέμα αυτό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Τίθενται τα ερωτήματα, προχωρεί κάποια συζήτηση για το τι θα γίνουν αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εύστοχε ερωτήσει, κυρία Ανδρίασεν και μετά κυρία Γκρέσλε. Κυρία... Ξέρω από την κυρία Γκρέσλε υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο, κυρία Ανδρίασεν. Thank you, Το μικρόφωνο της κυρίας Ανδρέασεν έχει ένα πρόβλημα. Το μικρόφωνο της κυρίας Ανδρέασεν έχει ένα πρόβλημα. Yeah. Ε, Απλώς θέλω να επισημάνω, για να απαντήσω κύριο, στα σχόλια του κύριου Φιέλνερ, ότι ανεξαρτήτως μεγέθους η υπηρεσία για την οποία μιλούμε είναι ένα όργανο που έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την κοινωνία. Άρα πρέπει να είναι αμέμπτου συμπεριφορά. Το να την συγχωνεύσουμε μέσα σε μια άλλη ε, ομάδα, οργανισμό κτλ. δεν αποτελεί λύση γιατί μάλλον θα επιμολύνει και την άλλη υπηρεσία παρά θα λύσει τα προβλήματα. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσα έχει. Ή απλώς να την κλείσουμε. Που ήταν η δική μου πρόταση. Πρέπει να είναι άμεμπτη η συμπεριφορά της για πόδος λογαριασμών. Αυτό πρέπει να πάντα να το έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ναι, ευχαριστώ. Με πρόλαβε ο κύριο Γκαέρ σε μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αποκεντρωμένε υπηρεσίε ε, εξασφαλίζουν τον προπολογισμό του μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν τον εισπράττουν απευθεία. Του τον χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα με κάποιο τρόπο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει. Έτσι δεν μπορεί να τους δίνει πάρτε τα χρήματα, κάντε τα ό,τι θέλετε και μετά το κοινοβούλιο θα πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ω εκ τούτου θα πρέπει να έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Και αυτή είναι η δουλειά την οποία έχουμε αναλάβει η κυρία Ριβελίνη και εγώ. Η υποχρέωση απόδοση λογαριασμών λοιπόν για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ακόμη και όταν υπάρχει ανάθεση για την εκτέλεση του προπολογισμού, δεν απαλλάσσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την υποχρέωση λογοδεσίας. Αυτό το βλέπουμε και στην απαλλαγή. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα δηλαδή. Να περιπέσουμε στην κατάσταση την ε, στρεβλή που βλέπουμε τώρα, ότι δηλαδή δεν είναι κανεί τελικά υπεύθυνο για λογοδοσία. Και εδώ πέρα θέλουμε συγκεκριμένε απαντήσεις. Κύριος, ε, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ο κύριος Γκρέι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν δεν απατώμε και ο κύριος Μαρίνη που είναι παρόν θα θέλει να λάβει το λόγο. Κύριε Γκρέι παρακαλώ εσείς πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πράγματι εξέτασε τις δραστηριότητες της ΣΕΠΟΛ πρώτα το Σεπτέμβριο του 2010. Τότε λοιπόν συντάξαμε μία έκθεση για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δράσης και για το κατά πόσο λήφθησαν υπόψη οι συστάσεις της Επιτροπής Επιλογής. Είχαν αναφερθεί 44 ορόσημα συσταγωγικά και αυτό το πρόγραμμα ε, δράσης ήταν ικανοποιητικό. 19 είχαν ολοκληρωθεί, 7 περίμεναν, 18 έτρεχαν ε, από τα ορόσημα πάντα. Ε, αυτά που δεν είχαν ολοκληρωθεί, η λυθυπόψη ήταν έτσι αμεληταία. Και Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα επανήλθαμε για να δούμε κατά πόσον η ΣΥΠΟΛ εφάρμοζε τις δικές μας τις συστάσεις. Γιατί εμείς ε, καταθέσαμε μια σειρά συστάσεων με βάση τα πορίσματά μας. Έξι λοιπόν είχαν εφαρμοστεί, δύο έτρεχαν και κάθε σύσταση είχε ορόσημα και τα ορόσημα είχαν ληφθεί υπόψη. Άρα δηλαδή σε γενικές γραμμές ήμασταν ικανοποιημένοι. Κρίναμε ότι το πρόγραμμα δράσεις ε, έχριζε διευκρινήσεων ε, σε αρκετά σημεία. Αυτές ήταν και οι ανησυχίες και επιφυλάξεις της ε, Επιτροπής της Αρχής Απαλλαγής. Εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και θα επανέλθουμε του χρόνου. Όσον αφορά τις γενικότερες επιφυλάξεις, πράγματι έχετε δίκιο. Πρόκειται για μια μικρή υπηρεσία που έχει ένα νέο ε, διευθυντή. Ε, τα νότητα στελέχη έχουν σχεδόν ανανεωθεί στο σύνολό τους. Άρα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια νεοσυσταθής υπηρεσία το 2008. Και εφόσον πρόκειται για μια μικρή υπηρεσία, το είπαν και ορισμένοι στην Επιτροπή, ε, πρέπει παρόλα αυτά αυτοί να σέβεται τους κανόνες Μπορεί κανείς να θέσει θέματα αποτελεσματικότητας ε, όταν μιλάμε για 25 υπαλλήλους και η ε, Κομισιόν από κοινού το Κοινοβούλιο πρέπει γενικότερα να εξετάσει το θέμα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι μικρές υπηρεσίες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν το στόχο τους ε, χωρίς όμως να υπάρχει επικάλυψη δομών με τις μεγάλες υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ομάδα εργασίας ε, και συνεχίζει τις εργασίες της. Ρωτήσατε κατόπιν ε, ποιο μάθημα μαθαίνει κανείς από τη ΣΥΠΟΛ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη δουλειά την ξεκινήσαμε το 2008. Στην πρώτη μας αποστολή εντοπίσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και μετά τα επισημάναμε στον τότε Διευθυντή ε, και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, σημειώθηκε κατόπιν πρόοδος στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πάμε πάλι στο θέμα της αποτελεσματικότητας. Ε, μπορεί κανείς να ε, διαφοροποιήσει τους δύο ρόλους της ΥΠΟΛ. Η ΥΠΟΛ ε, προσφέρει εκπαίδευση στους αστυνομικούς, αλλά εκείνος εκείνο που συζητήσαμε επίσης είναι ότι θα μπορούσε να είναι η γραμματεία για τέτοιου είδου δραστηριότητε που θα αναλάβει κάποιο άλλο φορέ. Νομίζω αυτά τα θέματα εξετάζει αυτή η διοργανική ομάδα εργασία. Τώρα, το τι κάνει η Κομισιόν για τέτοιου είδου θέματα. Ε, πρώτον, οι ρυθμιστικέ αρχές δεν είναι εκτελεστικές αρχές. Για να είναι εκτελεστικές αρχές, εκεί η Κομισιόν έχει εξουσία. Στις ρυθμιστικέ όμως δεν έχει. αυτέ συστήνονται μετά από πρόταση της Κομισιόν και η Κομισιόν έχει κατά κανόνα μία ψήφο στην ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι λίγο ε, γιατί έχουμε άλλους 27 που ψηφίζουν. Βεβαίω, η ε, Κομισιόν δίνει δάνεια και κατόπιν τούτου η υπηρεσία αυτή όπως και όλες οι άλλες πρέπει να σέβονται τους ε, όρους χορήγησης δανείου. Έχουμε δηλαδή αν θέλετε ε, κάποιες δυνατότητες σε πέντρο νομοθεσία για να ελέγχουμε την υπηρεσία ακόμα και να έχει μικρό διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα το επιβεβαιώσει ο συνάδελφός μου. Μόλις ενημερωθήκαμε αντί να δώσουμε στην υπηρεσία ε, τα ε, χρήματα σε ρευστό αρχίσαμε να πληρώνουμε με δόσεις και κάθε δόση ήταν συνάρτηση του κατά πόσον η υπηρεσία μπορούσε να μας αποδείξει ότι λάμβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι η Κομισιόν αντράνησε. Έγιναν ε, πολλές εκθέσεις από φορείς JLS για να ε, δούμε και να επηρεάσουμε ε, τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία αυτή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Πρόεδρε, υποστηρίζουμε και παρακολουθούμε την λειτουργία της ε, ΣΕΠΟΛ από τη θέσπιση της με στόχο να εξασφαλίσουμε την τήρηση των όρων του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, μη, ε, είναι μέλος μάλλον χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως, ε, οποτεδήποτε διαπιστώθηκαν αδυναμίες από τις ελεγκτικές αρχές, Φερρυπίν Ελές ζήτησε από τον προηγούμενο διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας μέσω επιστολής καλώντας τον να προσαρθεί στις Βρυξέλλες, να ε, συμμορφωθεί προς τις ε, οδηγίες των ελεγκτικών αρχών με βάση τους όρους που έχει προσδιορίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Και από το Μάρτιο του 2008 και ύστερα από τις προκαταρκτικές επιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ύστερα από επισκεψή του επιτόπου με την αυτοψία δηλαδή ε, που σχετίζεται με τον προπολογισμό 2007 συγκεκριμένα, Ύστερα λοιπόν από αυτή την προκατακτική διαπίστωση που οδήγησε σε πολλές ανησυχίες καθώς και να κάνει με προβλήματα ως προστιωτικές ε, δαπάνες, ε, ζητήματα φορολογικά κτλ. Η GTLS έστειλε ε, επιστολή και στην Όλαφ και έτσι ξεκίνησε η σχετική έρευνα της υπόθεσης. Ύστερα από αυτή την τεχνική λοιπόν, τεχνικού τύπου πρωτοβουλία, ξεκινούμε και μια πολιτική πρωτοβουλία το 2008 συγκεκριμένα στο πρώτο, και στο πρώτο ήμιση του 2009, την οποία στήριξε και η Τσεχική Προεδρία ιδιαίτερως. Το 2009 λοιπόν, κατόπιν αυτών των δρόσεων, οδηγήθηκε σε παρέτηση ο πρώην διευθυντής. Το Μάιο του 2009, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, Και εδώ σημειώνω ότι προβλήματα που είχαν εντοπιστεί το 2008 δεν βλέπουμε να επαναλαμβάνονται καθιονδήποτε τρόπο το 2009 ή με οποιαδήποτε μορφή. Για να σε εξηγήσω με παραδείγματα. Η αποτελεσματικότητα στη χρήση του προπολογισμού αυξήθηκε στο 47% από το 27% το 2009 σχέση με το 2008. Και όπως σωστά επενθύμησε ο κύριος Γκρέι νωρίτερα, παρακολουθούμε και τις ε, πληρωμές ε, από τον προπολογισμό στην ε, αποκεντρωμένη υπηρεσία και καταβάλαμε τα ποσά μόνο εκείνα τα οποία ήταν σύμφωνα με συγκεκριμένες θέσεις ρευστότητας και με συγκεκριμένες προβλέψεις έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο κατάχρησης επί του προπολογισμού. Ύστερα λοιπόν από την αλλαγή των διευθυντικών στελεχών πρέπει να πω ότι έχει ξεκινήσει μια νέα και πολύ υποσχόμενη φάση η Αστυνομική Ακαδημία. Όπως ήδη υπογραμμίστηκε η νέα διοίκηση καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να εξεύρει στα έκρημη ζητήματα. Ε, ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τι προσπάθειε τη Αστυνομική Ακαδημία για την επίλυση των υφισταμένων προβλημάτων και την εξασφάλιση των πολλαπλών μέσων που θα χρειαστούν για την ορθή λειτουργία τη και την παροχή τη υπηρεσία κατάρτιση αστυνομικών στελεχών. Επίση, συζητούμε μέσα σε μια ιστορική ομάδα εργασία την αναθεώρηση τη λειτουργία όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίε και να ενισχυθούν βέβαια τα σημεία μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βεβαίω του ελέγχου. Όσο δεν αφορά την αστυνομική ακαδημία έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία τη ε, αστυνομική ακαδημία, τη αποκεντρωμένη αυτή υπηρεσία, δηλαδή μέσω νομική βάση κτλ. Και Στόχος μας είναι να έχουμε μια αποτελεσματική υπηρεσία η οποία θα προσφέρει αποτελεσματική κατάρτιση αστυνομικών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Όση, έχετε κάποια παρατήρηση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι ενώπιόν σας από τότε που διορίστηκα να υπηρετήσω στο ελεγκτικό συνέδριο τον Απρίλιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, Πολλά εσωτερικά θέματα διαχείρισης έχουν αναφερθεί, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα ελέγχου που αναφέρθηκαν σήμερα. Ο δόκτωρ Μπάμφη και οι συνάδελφοί του έχουν ε, αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα που ήταν αντικείμενα επικρίσεων κατά σειρά ετών από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου. Καταρχήν, με χαρά ακούσαμε ότι ο εξωτερικός έλεγχος για τις ε, την κακοδιαχείριση και την ε, λανθασμένη ανάκτηση ήταν, ε, ναι, αντιμετωπίστηκε. Ήταν ένα θέμα το οποίο έχουμε επιστήσει την προσοχή εδώ και χρόνια. Επίσης το θέμα των συμβούλων ήταν προβληματικό εδώ και χρόνια. Δύο θέματα προκύπτουν από το πολιετές πρόγραμμα δράσης που έχει εισάγει η ΣΕΠΟΛ. Το ένα είναι ο διορισμός ενός λογιστή και επίσης ο διορισμός ενός ε, υπευθύνου για τις προμήθειες. Θα γνωρίζετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είχε επικρίνει την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΣΕΠΟΛ το 2007 και το 2008. Επίσης είχαμε κάποιες ε, επικρίσεις ε, για το, στην έκθεση την ελεγκτική του 2009. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια μικρή, ένας μικρός οργανισμός και το να διορθωθούν προβλήματα δημοσιονομικά το αυτό που χρειάζεται είναι ένας πολύ καλός λογιστής και ένα πολύ καλό ε, δημοσιονομικό πρόγραμμα και αυτό είναι ανακούφιση το να δούμε δηλαδή ότι σε ΣΕΠΟΛ πράγματι έχει ε, ε, προσλάβει έναν ειδικό λογιστή για αυτό το σκοπό. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, το ελεκτικό συνέδριο γνωρίζει το ρόλο του, ότι δηλαδή πρέπει να ελέγξει και τα θέματα αποτελεσματικότητας, αλλά και τα θέματα απόδοσης. Εμείς φροντίζουμε ώστε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να ε, δαπανώνται από αυτούς οι οποίοι ε, έχουν αναλάβει τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Στο πρόγραμμα εργασίας μας η δημοσίευση μιας έκθεσης για το, η σύγκριση του κόστους των ε, 22 οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα εξετάσουμε το κόστος ε, ως προς την αποτελεσματικότητα και την απόδοση ε, ώστε να προβούμε μετά σε αξιόπιστες ε, συστάσεις θα ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε χωρίς τις κατάλληλες αποδείξεις να πούμε αν η πόλη στη σημερινή της μορφή θα έχει μέλλον, αλλά ελπίζουμε όπως είπε και ο κύριος Γκρέι πως η έκθεσή μας θα ληφθεί υπόψη από εσά και του συναδέλφου σας σε σχέση με την ανάλυση αυτών των σημαντικών θεμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ματιέ, έχετε το λόγο. Ελπίζω κάπως να προχωρήσατε ως εισηγήτρια μετά όσα ακούσατε σήμερα. Θέλετε να ολοκληρώσετε με κάποια συμπεράσματα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι ο ίστατος έλεγχος πλέον. Βλέπω πως ο νέος διευθυντής, αλλά αυτό δεν είναι έκπληξη, το γνωρίζαμε, κληρονόμησε κάτι δυο ευχάριστο, είναι μια πραγματική πρόκληση και προσπαθώντας να βελτιώσει την κατάσταση από την στιγμή που έφτασε στην ΣΕΠΟΛ, Βεβαίως ε, όλα αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση με όλες του τις δυνάμεις. Σε σχέση με το Δικητικό Συμβούλιο, το τι συνέβη και γιατί το Δικητικό Συμβούλιο δεν αντέδρασε Πιστεύω πως δύο χρόνια χρειάστηκαν για να καταλάβουν ότι ο Διευθυντής δεν ήταν αποτελεσματικός και δεν μπορούσε να τηρήσει τους κανόνες, τους δημοσιονομικούς. Νομίζω πως είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, είναι μια συνολική ευθύνη την οποία δεν ανέλαβε κανείς. Σε πάση περιπτώσει τώρα ότι έγινε έγινε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λυπούμε που η Κομισιόν που επίσης ε, συμμετέχει στο δικαιωτικό Συμβούλιο δεν έχει περισσότερη εξουσία γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στο Διοικητικό Συμβούλιο που μπορούν να πούνε στο Διοικητικό Συμβούλιο τέρμα, τώρα τελείωσε αυτή η υπόθεση και τα 27 μέλη που έχουμε τώρα επιτέλους στον κατάλογο των ονομάτων, επιτέλους δεν τον έχω τον κατάλογο εδώ και πολύ καιρό, αλλά επιτέλους τον έχω στη διάθεσή μου, αλλά τελικά για διάφορους, για πολλούς και διάφορους λόγους, ίσως και για πολιτικούς μόνο λόγους, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Και πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν η Κομισιόν είχε δικαίωμα ψήφου, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοια προβλήματα όπως αυτά που φτάσαμε στη ΣΕΠΟΛ. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Τώρα βέβαια θα πρέπει να κλείσουν κάποια στιγμή οι λογαριασμοί γιατί έχουμε μπει στη διαδικασία απαλλαγής για το 2009 και πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούμε δηλαδή επαόριστον να καθυστερούμε αυτή την υπόθεση για όλα τα μέρη και για την εισηγήτρια, ε, πρέπει να σας το πω και αυτό. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε στο κλείσιμο των λογαριασμών, εκτός και αν κάποιος συνάδελφος είναι αντίθετος. Τώρα βέβαια εσείς πρόεδρε θα πρέπει να λάβετε την απόφαση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, προβλέπετε το κλείσιμο αυτών των οργανισμών για την Πέμπτη. Και μπορούμε να διαβιβάσουμε το ντοσέ, το ντοσιέ, τον κύριο Σταυρακάκη που είναι ο εισηγητής για την απαλλαγή 2009. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία με αυτή την υπόθεση όπως και εμείς κύριε Σταυρακάκη διότι τόσο ο πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο διευθυντής της ΕΠΟΛ να μπορούν να έρχονται ε, εδώ ευχαρίστως χωρίς να φοβούνται μήπως συναντήσουν κανέναν από την ε, Κουκομπού ή τη Λίμπε. Αυτά. Πέρα τη υπόθεση, ε, περνάμε στο σημείο 5, την έκθεση Κέστιγκερ. Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 10 του 2010 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου. En geschreven door ehm, Hubert Weber, lid van de Rekenkamer, en zijn eh, medewerkers θα καλέσω τον κύριο Βέμπερ να μας ε, κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις στην εισήγηση και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Κέστιγκερ να μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας σας. Ο κύριος Κέστιγκερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτή την ε, έκθεση σχετικά με τα ιδιαίτερα μέτρα που ελήφθησαν προς όφελος της Γεωργίας στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Τα ειδικά αυτά μέτρα ελήφθησαν το 2006 με στόχο να υποβληθούν στην Κομισιόν έτσι ώστε η Κομισιόν ε, να προβλέψει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών τόσο κατά την αποκέντρωση όσο και ε, κατά την ε, λήψη αποφάσεων. Το, το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν διαπιστώνει ότι αυτά τα μέτρα κατά το μάλλον ήταν, είχαν σημαντικές προεκτάσεις στη γεωργία αυτών των ε, περιοχών. Βέβαια ε, διαπιστώθηκαν και αρκετές αδυναμίες που σημαίνει ότι εδώ πράγματι είναι δυνατόν να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις για να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα των μέτρων. Είχαμε κατόπιν την μεταρρύθμιση του 2006, η οποία ε, μεταρρύθμιση αυτή επικεντρώνεται στην αποκέντρωση. Τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες. Και η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να ελέγχεται η συμβατότητα και η συνοχή των προγραμμάτων χωρίς βέβαια να θέλει η ίδια να συμβάλλει σε θέματα διαχείρισης και κατάρτισης των προγραμμάτων. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των και την εκτέλεση των προγραμμάτων, το λεκτικό συνέδριο εντόπισε μέτρα ή αν θέλετε και δράσεις που δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Αυτές οι δράσεις. Ε, εξάλλου, επειδή τα μέτρα ε, είναι και πολύ περίπλοκα, δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή επιμένει τα μέτρα να αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια. Βέβαια αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο. Οι εκθέσεις εφαρμογής που συντάσσονται από την Επιτροπή κάθε χρόνο δεν είναι ομοιόμορφες οι εκθέσεις αυτές, αλλά ούτε και πλήρεις και γι' αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κατόπιν τούτου, το ελεγκτικό συνέδριο έχει υποβάλει συστάσεις ε, οι οποίες θα επιτρέψουν τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαχείριση των ειδικών αυτών μέτρων. Οι συστάσεις λοιπόν αφορούν και, και αναφέρω πρώτον την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων ιδιαίτερα η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνουν τα κρατημέλη για το ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι και να τους δίνει και ένα ενιαίο πλαίσιο δικτών απόδυσης. Δεύτερον, την αναθεώρηση της καταληκτικής προθεσμίας ε, για την υποβολή και την ε, δρομολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Τρίτον, την τροποποίηση των μέτρων όπου εντοπίστηκαν ε, αδυναμίες ε, τα μέτρα αυτά πρέπει να κυρίως από την Κομισιόν. Και τέλος, τη διασφάλιση ε, διαδικασιών ελέγχου, ε, τα οποία, οι οποίοι έλεγχοι θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στα μέτρα που θα έχουν ληφθεί. Σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κύριε Βίμπα. Ευχαριστούμε για τις εξηγήσει μας δώσετε η κυρία Κιώστιγκα που σας παρακολούθησε. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Κυρία Κιώστιγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ελεγκτικό συνέδριο για αυτά τα ιδιαίτερα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστώ ε, κυρίως τον κύριο Βίμπερ αυτό ήταν αρμόδιος από το Λεγκτικό Συνέδριο ε, για τη συνεργασία μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα ιδιαίτερα μέτρα έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ε, ενσωμάτωση. Ε, το 83 μέχρι το 88 εφαρμόστηκαν προγράμματα και το 2006 υπήρξε μεταρρύθμιση των προγραμμάτων για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Στο πλαίσιο λοιπόν των προγραμμάτων που κατέθηκαν ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις. Πρώτον, να μην επιβάλλονται δασμοί σε εισαγωγέ από τρίτε χώρε ή αν θέλετε επιδότηση για προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και δεύτερον, να υπάρξει περαιτέρω αξιολόγηση, ε, μάλλον εξέλιξη των, της γεωργίας, ε, της γεωργικής παραγωγής με επιδοτήσεις, με πριμ και με άλλες μορφές πληρωμών. Ε, το χρονικό διάστημα από το 2007 μέχρι το 2010 που έλεγξε το ελεκτικό συνέδριο αφορούσαν 1,6 περίπου δις ευρώ. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν έλεγξε την αποτελεσματικότητα των μέτρων από τη μεταρρύθμιση του 2006 κυρίως ε, τα προγράμματα ε, που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων αλλά και στον έλεγχο των μέτρων. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου τις οποίες και στηρίζω. Πρώτα απ' όλα θα αναφέρω τέσσερα σημεία, τα οποία κατά άποψή μου είναι μεγάλη σημασία. Πρώτον, δείκτες ελέγχου χαιρετίζω τις διαβουλεύσεις της Κομισιόν με τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη σχετικά με τους δείκτες ελέγχου που θα πρέπει να ισχύουν από το 2011. Εδώ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία έτσι ώστε για όλα τα προγράμματα να υπάρχουν ενιαίοι δείκτες ελέγχου. Δεύτερο σημείο αφορά τον τομέα των εφάπαξ ποσών. Ε, τα εφάπαξ αυτά ποσά ε, για την παραγωγή αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Κατανοώ βέβαια ότι σε ορισμένες περιοχές είναι απαραίτητο να δίδονται ε, κάποια εφάπαξ ποσά όμως τα ποσά αυτά πολύ συχνά ε, βρίσκονται σε αντίφαση με την αηφόρο ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό είναι και το διάστημα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτή τη στιγμή γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Η Κομισιόν προτείνει να αξιολογούνται τα προγράμματα κάθε τρία χρόνια και το ελεγκτικό συνέδριο κάθε χρόνο. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ε, εδώ για να καταλήξει κανείς κάπου θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξή στοιχεία. Αν γίνεται η αξιολόγηση κάθε χρόνο, δεν μπορεί να υπάρξει εμβριθής ανάλυση των προγραμμάτων. Ε, θα πρόκειται περισσότερο για μια επανεξέταση η οποία μεταξύ άλλων θα διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα κράτη-μέλη πράγματι αξιολογούνται και δεν εξαφανίζονται σε κάποιο ντουλάπι. Η ε, Κομισιόν έχει ε, προτείνει συγκεκριμένες ε, απόψεις επί του θέματος αυτού. Για να υπάρχει βέλτιστη αξιολόγηση ε, θα πρέπει βεβαίως να υπήρχε και ένα σύστημα ενημέρωσης το οποίο θα βοηθούσε ε, στο να υπάρχει καλύτερη συγκέντρωση των δεδομένων και καλύτερο έλεγχο ε, του input και του output. Το τελευταίο θέμα που θέλω να φέρω αφορά την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει σημαντικό ρόλο κατά την υποστήριξη ε, των κρατών μελών. Η Κομισιόν πρέπει να εξετάσει το κατά πόσο τα προγράμματα είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο. Από την άλλη όμω πρέπει να υπάρχει και κάποιο συντονισμό που πρέπει να τον διασφαλίζει η Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και στις διαβουλεύσεις ε, για την ε, θέσπιση κοινών δικτών. Εγώ στηρίζω την προσέγγιση της ε, Κομισιόν και θα ήθελα, παραθέτω μάλλον τα εξή. Καλούνται τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν μέτρα για την μέτρηση των προγραμμάτων. Κάτι τέτοιο λείπει μέχρι τώρα. Τέλο παράθεση. Εδώ λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί εκείνο που μπορεί να γίνει σε μικρό επίπεδο, δηλαδή σε τέσσερα κράτη-μέλη, προφανώ μπορεί να χρησιμοποιήσει και για άλλου τομεί χρηματοδότηση. Τελειώνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι 16 από του 24 τομεί που ελέγχθηκαν ε, παρουσίασαν παρουσίασαν ε, σημαντικά βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Πέραν αυτού, τα ειδικά αυτά μέτρα οδήγησαν στη βελτίωση του εισοδήματος ε, των γεωργών και στην διατήρηση της γεωργίας. Άρα δηλαδή τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε αυτές τις περιοχές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίζονται κυρίως, διασφαλίζονται τα προστοζήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεση που υπέβαλε και περιμένουμε μεγάλη χαρά ερωτήσεις που τυχόν έχουν οι συνάδελφοι πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Όχι, τότε στρέφαμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροφή. Το πει. Κύριος Μποσάχ. Και συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω το όνομά σας. Θέλει να λάβει το λόγο. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει απαντήσεις στα όσα ακούστηκαν, γιατί κατόπιν των ε, συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου είχα την εντύπωση που ήσασταν μάλλον θετική στις προτάσεις αυτές. Δεν είναι μόνο σαφές ε, όταν βλέπουμε τροπολογίες για κάποιον ε, κανονισμό, εάν δίνετε κάποιες συνέχεια από πλευρά σας. Έχετε λοιπόν κάνει προτάσεις ή σκοπεύετε να καταθέσετε τέτοιου είδου προτάσει αυτά ως συμπληρωματική ερώτηση για τον κύριο Μποσόρτ. Κύριε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή, καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά την κυρία Κέστιγκερ για τις προτάσει και συστάσεις. Είναι πολύ αξιόλογη, πολύ αξιόλογη συμβολή στην ε, ενεξελίξη τώρα επανεξέταση του κανονισμού του σχετικού με τις εξόχους από περιοχές και τα μικρά νησιά ε, στην οποία προβαίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά θα λάβει υπόψη τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στον κανονισμό που θα καταθέσει ω προ τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στι εξόχω απομακρυσμένε περιοχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει λοιπόν δουλειά εν εξελίξη και οι συστάσει αυτέ θα ενσωματωθούν στην, ε, στο δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερως ότι το άρθρο 20 349 ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ρητά πως συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή των αξιόχως απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, παραγωγή και την ε, προμήθεια σε υλικό και τα απαραίτητα των περιοχών αυτών θα λαμβάνεται με συγκεκριμένες δράσεις. Τα προγράμματα λοιπόν αυτά ε, έτυχαν να θεωρήσω στο 2006 και με στόχο, όπως είπε και ο κύριος Βέιμπερ πολύ σωστά, ένα υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας στη χείρισή τους, ε, όσο πιο πολύ δηλαδή ε, αποκεντρωμένη διαχείριση και τα κράτη-μέλη κατέστησαν υπεύθυνα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εποπτεία των προγραμμάτων. Αυτό ήταν και κατά την άποψή μας ο καλύτερος τρόπος να βαθύνουμε στα προγράμματα αυτά και να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες στην κάθε περιφέρεια. Και τώρα λοιπόν με την ευκαιρία του ελέγχου ε, ε, αξιολογείται το, ο βαθμός στον οποίο αυτή η μεταρρύθμιση έχει προσφέρει περισσότερη ουσιαστική υποστήριξη στις εξόχω μαξιπέρας περιοχές και τα νησιά του Αιγαίου. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ξεκινώντας το άριστο πνεύμα συνεργασίας και την επικοδομητική προσέγγιση αυτής της ε, ελεγκτικής δράσης. Ελάχιστα τα σημεία διαφωνία σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου και μέσα από τις συστάσεις τις οποίες εν γέννη καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που και εσείς άλλωστε επισημάνατε, Πρόεδρε, θα αποτελέσουν καλή βάση για εξέλιξη της διαχείρισης του ΠΟΣΕΙ στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερω αισθάνεται ικανοποίηση προς τα, από τα συμπεράσματα μάλλον του ελεκτικού συνεδρίου για την ανάπτυξη οργίας στις εξοχώς αποκεντρωμένε περιοχές και τη, τα νησιά του Αιγαίου ότι είναι δηλαδή πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα για την ανάπτυξη οργίας στις εν περιοχές και όπω είπατε και εσεί, κύριε Βέβαιο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε απόλυτη ταύτιση απόψεων σε κάθε σημείο. Έχουν διατυπωθεί κάποιε διαφωνίε προ τι συστάσει. Έχει παρακολουθήσει και με τι προτάσει η κυρία Κέστιγκερ και πιστεύουμε ότι ίσω χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση ορισμένων σημείων σημείων. Θα μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ σε πέντε μόνο σημεία πολύ σύντομα. Πρώτον, όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τη βελτίωση τη εποπτεία και τη αποτελεσματικότητα, εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την στήριξη που προσφέρει η κυρία Κέστιγκερ στην έκθεση και τι μεταρρυθμίσει του 2006. Μεταθέτουμε δηλαδή την ευθύνη πλέον στα κράτη-μέλη για τον προσδιορισμό των προγραμμάτων και Είμαστε της απόψεως ότι συγκεκριμένα μέτρα ε, θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται ιδιαίτερε ανάγκε κάθε περιοχή. Αλλά ε, επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε, όπω άλλωστε και η κυρία Κρίστιν Κέρεν προκειμένου, ότι αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και βελτίωση τη τάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στην οποία σκοπεύουμε να προβούμε με του εξή δύο τρόπου. Πρώτον, Θέλουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τις απόψεις μας ως προς την μεταρρύθμιση του ΠΟΣΕΙ ε, που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και που σκοπεύουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τώρα. Πρόκειται για ένα πακέτο, για ένα σύνολο εργαλείων δηλαδή, ε, για την καλύτερη εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και στη συνέχεια έχουμε καταθέσει προτάσεις για έναν ενορμονισμένο πλαίσιο ε, κοινών δικτών για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των ε, προγραμμάτων κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτοί οι κοινοί δείκτες λοιπόν συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα πληροφορίες για την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερως ε, αλλαγές στην περιοχή, ζωικό κεφάλαιο, συγκομιδή, αλλά και στον πληθυσμό. Ιδιαίτερα δε ως προς την κατάσταση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, ή της απασχόλησης γενικότερα. Δεύτερη σύσταση. Διευκόλυνση ω προ την ετήσια διαδικασία αν των κρατών μελών, που αποτελεί επίση πολύ σημαντική σύσταση. Και πάλι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ακολουθήσει τις ε, συστάσεις και αυτό έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η ε, ετήσια διαδικασία. Και εδώ έχουμε δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, οι τροποποιήσεις που προτείνονται κάθε χρόνο από τα κράτη-μέλη να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς όμως να υπάρχει έγκριση μια τυπική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, με μια καλύτερη καθοδήγηση όλε αυτέ τις διαδικασίε, ναι. βελτιώνουμε τη ε, διαδικασία με τι τροποποιήσει, χωρί όμω να εμπλέκεται μια τυπική διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι κερδίζουμε χρόνο και για την προετοιμασία των τροποποιήσεων αυτών. Και εδώ έχουμε το δεύτερο στοιχείο τη εν λόγω συστάσεω, ότι για να ακολουθήσουμε τι προτάσει του ελεγκτικού συνεδρίου, θέλουμε να αναβάλουμε την προθεσμία, να παρατείνουμε δηλαδή την προθεσμία κατά την οποία μπορούν τα κράτη-μέλη να καταθέσουν τις τροποποίησεις τους. Κατά δύο μήνες, αντί για 1η ε, Αυγούστου, θα έχουμε καταληκτική προθεσμία την 21η Σεπτεμβρίου και έτσι τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευκαιρία και να προσδιορίζουν τις τροποποίησεις τους και να έρχονται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς και να κάνουν σχετική προπαρασκευή. Ε, η, δεύτερη, η τρίτη μάλλον πρόταση έχει να κάνει με την εμπλοκή των ενδιαφερομένων καλύτερη ανάλυση, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων. Και πάλι συμφωνεί εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την σημασία της εμπλοκής ε, των ε, ενδιαφερομένων φορέων και βεβαίως αν έχουμε αυτούς τους επιπλέον δύο μήνες θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη συμμετοχή στη δικασία των ε, φορέων αυτών ιδιαίτερα δεν έχουμε καταθέσει προτάσει προ τα κράτη-μέλη για μια πιο στρατηγική προσέγγιση κατά τον προσδιορισμό και υποβολή προτάσεων για τροποποίηση στα εν προγράμματα, κατά τρόπο πιο διαρθρωμένο δηλαδή, με περισσότερη στόχευση, καλύτερη στόχευση στο αποτέλεσμα και πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των αναγκών της κάθε περιφέρειας. Τέταρτη παρατήρηση. Κοινή ρυθμιστική δείκτες και αιτήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων. Αναφέρθηκε και από την κυρία Κωστινέρ και από τον κύριο Βέιμπερ ότι η πενταετία είναι υπερβολικά μακρά περίοδος, το ένα έτος είναι υπερβολικά σύντομη περίοδος και ως εκ τούτου. Εμείς φρονούμε ότι με μία προσέγγιση που θα στηρίζεται σε κοινού δείκτες και που θα ε, επιτρέπει κάθε χρόνο να γίνεται η εποπτεία, η παρακολούθηση, μπορούμε να έχουμε ένα καλό μέσον, ένα καλό εργαλείο να επιδιώκουμε την επανεστίαση όπου υπάρχει πρόβλημα ως προς τις ανάγκες. Και βεβαίως τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί στο στόχο αυτόν, οι δείκτες δηλαδή ισχύουν ήδη από εφέτος. Είναι ενισχύ οι δείκτες και προσφέρουν και μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όταν έχουμε να κάνουμε με την αξιολόγηση των, της εκθέσεως ως προς τις ελλείψεις της δηλαδή. Δεν πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπογραμμίσει το εξή ότι δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε εις βάθος σε αιτήσια βάση ολόκληρο ένα πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια πολυετή προσέγγιση για αυτή την αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή ορίζεται η περίοδος της πενταετίας, η περίοδος αναφοράς. Ε, αυτήν θα ακολουθήσουμε, αλλά θέλουμε βεβαίω και τι προσπάθειε μα να τι επικεντρώσουμε σε έναν ετήσιο εναρμονισμένο δείκτη. Μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή για ετήσιο εναρμονισμένο δείκτη. Και για να κλείσω, η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε στόχο έχει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Ναι, μεν, πλην όμω, πιστεύουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο ήταν, κάπως, ήταν μάλλον υπερβολικά αυστηρό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχουμε τακτικέ επαφέ με τις αρχές και στις εξόχως αποκεντρωμένες περιοχές και με τα, των, των κρατών μελών τις αρχές. Υπάρχει βεβαίω πολύ ακόμη πεδίο για καλύτερη συνεργασία. Ως ήθιστε η συνεργασία μπορεί πάντοτε να βελτιωθεί. Και η Επιτροπή σας δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για πιο στενή και κατά πάσα πιθανότητα και πιο θεσμοθετημένη συνεργασία στο βαθμό του δυνατού. Αλλά για να κάνω τελευταία μου και καταληκτική ε, παρατήρηση κατόπιν ε, των όσων ακούσαμε από τον κύριο Βέμπερ. Το ελεγκτικό συνεδρίο λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις τώρα κοιτάξατε όλα τα προγράμματα και τη θέσπιση των προγραμμάτων και θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι είναι σύνομα με τον κανονισμό και βλέπουμε ότι δεν έχετε ε, λάβει ενεργό μέρος στην διατύπωση των προτάσεων και την, ε, δεν έχετε παράσει συμβολές στα κράτη-μέλη για τη διατύπωση των προγραμμάτων και των σχεδίων. Όμως πρέπει εδώ να σαφέ ότι πρωταρχικό μας καθήκον και κύριο καθήκον μας είναι να βεβαιωνόμαστε ότι τα όσα γίνονται και οι δαπάνες βέβαια που προκύπτουν από αυτά τα προγράμματα είναι σύνομες με τον κανονισμό. με την μετάθεση των ε, ευθύνων για τα προγράμματα στα κράτη-μέλη, αυτά φέρουν την ευθύνη μεν, πλην όμως εμείς είμαστε στη διάθεσή τους για να τα ε, συνδράμουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Και φυσικά, στο βαθμό αυτό, λαμβάνουμε υπόψη τις παρατηρήσεις κυρία κυρίας Έτσι φτάνω στο τέλος των παρατηρήσεων και των σχολείων μου. Ευχαριστώ πολύ το ελεγκτικό συνέδριο και την κυρία Κέστιγκερ για την επικοδομητική προσέγγιση. Είμαστε στη θέση σας για... και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση εφόσον κρίνεται ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί αυτό το συστάσιο. Σας ευχαριστώ. Μετά τα όσα ακούσαμε, Δύο θέλω να παρέμβω, ο κύριος Γκέγερ και ο κύριος Μούλντερ. Ο κύριος Γκάγερ πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, ευχαριστώ την εισηγητρία και τον κύριο Βίμπα για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπαν. Άκουσα την άποψη της Κομισιόν και μου γεννήθηκαν ε, τρεις ερωτήσεις. Ίσως ε, να επηρεάστηκα από τις ε, διαφωνίες που έχουμε ή είχαμε τους τελευταίους μήνες με τους εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου για την κατάρτιση του προπολογισμού. Αλλά από αυτά που είπατε, έτσι σαν να κατάλαβα ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όσον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Εσείς τουλάχιστον δεν είστε ιδιαίτερα ευτυχείς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εσάς Κομισιόν, πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αν ναι πώς, δεύτερο ερώτημα. Αυτό που είπατε για το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών. Πολύ ωραία ιδέα. Εμένα, ε, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το εξής οι χώροι για τους οποίους μιλάμε, τα νησιά, αλλά και οι χώροι παραγωγής. Πώς είναι δυνατόν να γίνει εκεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Δηλαδή οι περιοχές αυτές είναι συγκρίσιμες και ανέ ναι, Και το τρίτο μου ερώτημα αφορά τον κύριο Βίμπα και το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή κατά τη δική σας άποψη θέλω να ξέρω ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ενσωμάτωση ε, είναι ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή τα κονδύλια χρησιμοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ή μήπως έχει να προτείνετε κάτι στην Κομισιόν. Αν μπορούσατε κύριε Βέμπερ να σχολέσετε και τις δύο ερωτήσεις που προηγήθηκαν θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τις ε, ιδιαίτερα απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα όσα ισχύουν στην κοινή γεωργική πολιτική, αλλά διάβασα στην έκθεση ότι μπορεί να αποφασίσουμε ότι αυτές να, εξερίζονται, να εξαιρούνται από την ε, ενιαία πληρωμή ή κατά αγρόκτημα ε, κατά εκμετάλλευση. Αλλά είναι κάπως ε, ε, εντυπωσιακό για μένα. Το σημείο 46 λέει ότι τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα μέτρα είναι γενικά πολύ μικρά. Η πληρωμή είναι 203 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, ενώ η συνηθέστερη πληρωμή ανέρχεται σε 58 ευρώ ετησίως. Αν ήμουν εγώ Γιώργος και λάμβανα 58 ευρώ ετησίω για να αυξήσω την ανταγωνιστικότητά μου και όλα τα άλλα στο νησί. Μα πώς το κάνω είναι αυτό δυνατόν <laughs> με ένα τέτοιο ποσό. Είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός ελέγχου και όλα τα συμπαραμαρτούντα όταν ο δικαιούχος ε, παίρνει όλα και όλα 60 ευρώ το χρόνο. Εγώ δεν νομίζω ότι αξίζει το κόπο. Μήπως κάνω λάθος αυτό το συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν για την Κομισιόν και τον κύριο Βέμπερ. Κομισιόν πρώτα. Δύο ερωτήσεις του κυρίου Γκέιερ και μία του κυρίου Μίλτερ. Επειδή η ερώτηση, η τέτοια στα γερμανικά θα μου επιτρέψει να απαντήσω και εγώ στα γερμανικά. Έχετε δίκιο κύριε Γκάια. Δηλαδή την αποτελεσματικότητα των κρατών μελών κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων ε, την αντιμετωπίζουμε πολύ κριτικά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Γιατί, διότι διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη μετά τη μεταρρύθμιση θέλησαν να, αφήσουν, να συνεχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα που είχαν ε, ήδη δρομολογηθεί και να κάνουν έτσι κάποιες εμβαλωματικές διορθώσεις. Ήταν λοιπόν μια επιλογή αυτή των ε, κρατών μελών ε, κάτι που προβλεπόταν στη μεταρρύθμιση. Το δικό μας όμως το καθήκον, και εδώ συμφωνούμε με κάποιες από τις συστάσεις, είναι να ε, φτάσουν τα κράτη-μέλη σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα από αυτήν την επιλογή και από εμβαλωματικές λύσεις να καταλήξουν σε μία ριζική αναθεώρηση και αν θέλετε και μία ε, αλλαγή μεγάλης κλίμακας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα πάντα. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επικρίνουμε δρυμύτατα τα κράτη-μέλη διότι και η εναλλαγή, μάλλον, η εναλλακτική λύση που ε, έχουν εμπλέξει τα κράτη-μέλη έχει γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα τις βέλτιστες ε, πρακτικές, πράγματι δίκιο έχετε. Οι περιοχές αυτές δεν είναι συγκρίσιμες, ε, ποικίλουν πολύ και δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Εκείνο όμως ε, που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αναλύσεις, γιατί υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Παραδείγματο χάρη, η μορφή των επιδοτήσεων. Ποια μορφή να επιλέξουμε, να επιλέξουμε τα καταποκοπή ποσά, ε, κάποια άλλη μορφή πληρωμών. Ε, αυτό μπορεί να ισχύσει για όλες τις περιοχές που σημαίνει δηλαδή εξετάζουμε τα θέματα σημείο προς σημείο για να καταλήξουμε πού είναι δυνατόν να επηρεάσουν οι βέλτιστες πρακτικές στις περιοχές και αν όχι όλες τις περιοχές, τουλάχιστον κάποιες. Αν υπάρχουν κάποια μέτρα που λειτουργούν σωστά, πρέπει να τα δημοσιοποιήσουμε και να διαδοθούν τα μέτρα αυτά και σε άλλες περιοχές. Αν θέλετε, αυτές είναι οι βέλτιστες ε, πρακτικές. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω αγγλικά. Για να απαντήσω στον κύριο Μούλντερ και στην τρίτη ερώτηση, έχετε δίκιο. Οι εξόχως περιοχέ περιοχές ε, έχουν βγει από το ε, SPS. Αλλά ο υπολογισμό είναι κάπω διαφορετικό γιατί υπάρχουν διάφορε πληρωμέ στι περιοχέ αυτέ. Έχουμε ένα βασικό πριμ που ήθιστε να είναι αποσυνδεδεμένο μέχρι μέση αξία 203 ευρώ. Έχετε τα top-ups και έχετε και ειδικέ πληρωμέ. Πρέπει δηλαδή να δει κανεί το τελικό ποσό που παίρνει ο Γιώργο. Ο Γιώργο δεν παίρνει μονάχα αυτό το ποσό. Είναι ε, διάφορες πηγές χρηματοδότησης από συνδεδεμένες, συνδεδεμένες, εθνικά top-ups και όλα αυτά είναι τμήμα της τελικής πληρωμής που τελικά λαμβάνει ο δικαιούχος. Παραμένει βεβαίως το ερώτημα ακόμα και αν δεν είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του εισοδήματος του Γεωργού, γιατί να προβλεφθεί ένα ολόκληρο σύστημα για να ελεγχθούν 58 ευρώ ετησίως. Ο κύριος Μιλτερ είναι ειδικό της ε, Γεωργίας. Κύριε Βέμπερ, θέλετε να απαντήσετε στην τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Λάιπ μίλησε για τον ιδεατό κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως και στον ιδεατό κόσμο μπορούν να υπάρξουν ε, βελτιώσεις. Το ίδιο ισχύει και εδώ με την μεταρρύθμιση ΠΟΣΕΙ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν τελικά ε, δεχθούμε τις ε, συστάσεις θα επιτύχουμε βελτιώσεις. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι άλλο. Όσον αφορά τη Γεωργία, εγώ ίδιος συμμετείχα στους ελέγχους που έγιναν στοιχείο στην Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι κατ' ουσίαν μιλάμε για μικρούτσικες, πολύ πολύ μικρές ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ε, αγωνίζονται να παραμείνουν ζωή, αγωνίζονται να διατηρήσουν τους ελαιώνες. Και ξέρετε, ακόμα και τα 80 ευρώ, αν θέλετε, για τους ανθρώπους αυτούς είναι πάρα πολλά χρήματα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κέστιγκερ, για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βέιμπερ και τον κύριο Μπόχαρτ. Ε, ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που έδωσαν, για τις ε, ξεκάθαρες απαντήσεις. Ευχαριστώ επίσης ε, και τους ε, συναδέλφους για τις προτάσεις που κατέθεσαν. Νομίζω όλοι συμφωνούμε Συμφωνεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω, να επανεξεταστούν και ε, τα μέτρα να ληφθούν οποτεδήποτε είναι απαραίτητα. Έτσι λοιπόν οι προτάσεις που ανέφερε η Κομισιόν σχετικά με την ε, αξιολόγηση σε αιτήσια βάση, αυτή η πρόταση ε, μου φάνηκε σωστή, θα τη σκεφτώ και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη που είχαμε προβλέψει για σήμερα. Αύριο θα ξεκινήσουμε στις 9 το πρωί. Θα έχουμε μεταξύ μας την Κάθριν Ντέι, Γενική Γραμματέα της Κομισιόν. Μπορέσαμε να δουλέψουμε πολύ ωραία σήμερα. Έδωσα το λόγο άπλυτα σε όλους. Φοβούμαι πως αύριο θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα γιατί θα είναι πιο φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό και καλό όλους τους συναδέλφους να είναι εδώ ακριβώς στις 9 ώστε να ξεκινήσουμε χωρίς καμία καθυστέρηση στην αυριανή συνεδρίαση με την παρουσία της κυρίας Ντέι.